Καθίστε παρακαλώ. Ο συνάδελφος θα πάρει το λόγο. Eh, λοιπόν, ε, θα αναλάβω εγώ την ε, Προεδρία γιατί ο κύριος Ντεμάγιστρης έρχεται γιατί μόλις προσγειώθηκε από την Ιταλία και ε, μόλις έφτασε στις Βρυξέλλες. Ε, αυτό είναι το, το οικολογικό αποτύπωμα που αφήνουμε. Ας ρίξουμε μια ματιά προτείνω στην ημερήσια διάταξη την οποία ούτως ή άλλως ε, θα πρέπει να ανατρέψουμε γιατί στο σημείο 11 την έκθεση Κοτσολίνο για προστασία των οικονομικών σφαιρών της κενότητας ε, η έκθεση του 2008 πρέπει να φύγει ο εισηγητής 11 ε, η ώρα από ό,τι κατάλαβα οπότε προτείνω γιατί έχουμε και ραντεβού με τους δύο επιτρόπους, τον κύριο, τον κύριο Κάλλας και τον κύριο Σεμέτα. Οπότε προτείνω να δούμε πρώτα την έκθεση Κοτσολίνο και μετά να ακούσουμε τον ε, κύριο Κάλας. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή της ημερήσιας ε, διάταξης, την οποία προτείνω και η δεύτερη αλλαγή είναι ένα σημείο το οποίο προέκυψε αυτή τη βδομάδα και στην συνεδρίαση των συντονιστών και στην προηγούμενη συνεδρίαση το γεγονός πως ε, αναμένουμε μία έκθεση ή εν πάση περιπτώσει μία ενημέρωση από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Όλαφ καθώς προέκυψαν κάποιες δυσκολίες και ζητήσαμε μία νομική γνωμοδότηση από την υπηρεσία μας και με πρόταση της κυρίας Γκρέσλε, η οποία είναι η συντονίστρια της ε, μεγαλύτερης ομάδας του Κοινοβουλίου του ΕΛΚ, δηλαδή προτείνω να δούμε αυτό το σημείο πρώτο-πρώτο, γιατί Πρέπει να γνωρίζουμε αυτό το θέμα πριν γίνει η συζήτηση με τους κυρίους ε, Σεμέτα και Κάλες για να μπορέσουμε να συζητήσουμε σε μια πιο λογική βάση. Οπότε αυτές είναι οι αλλαγές. Πρώτα απ' όλα δηλαδή να ακούσουμε την ε, νομική υπηρεσία, μετά να μιλήσουμε με τον κύριο Σεμέτα μία ώρα, μετά την έκθεση Κοτσολίνο και μετά να μιλήσουμε άλλη μία ώρα με τον κύριο Κάλλας. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο προτείνουμε. Συμφωνείτε με αυτή την αλλαγή της ημερήσιας διάταξης. Ναι, ωραία, ευχαριστώ. Οπότε απευθύνομαι τώρα στην νομική υπηρεσία να μας ενημερώσει για την κρίση της, για το που κατέληξε όσον αφορά αυτόν τον διορισμό. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα αγγλικά καθώς αυτή τη γλώσσα είναι και η γνωμοδότησή μας. σχετικά με την ενδιάμεση διαδοχή του κυρίου Μπρούνερ του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ έχετε λάβει την επιστολή του Αντιπρόεδρου Κάλλας η οποία λέγει ότι στην περίπτωση του θανάτου του Γενικού Διευθυντή, αυτός ο οποίος διορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τον αντικαταστήσει, για να τον αντικαταστήσει, αντικαθιστά ταυτόχρονα και τον Γενικό Διευθυντή. Αυτό βασίζεται στο άρθρο 27 του κανονισμού λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέγεται εκεί όταν εμποδίζεται από το να λειτουργήσει ο Γενικός Διευθυντής, σε αυτή την περίπτωση ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει την υπηρεσία αυτή ή κάποιος άλλος ο οποίος ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια τακτική θα λέγαμε αντικατάσταση ενός τακτικού γενικού διευθυντού. Εμείς διαφωνούμε σε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για μια τακτική αντικατάσταση. Δεν αντικαθίσταται κάποιος επειδή είναι απόν. Εδώ γνωρίζουμε ότι αποδίωσε ο συγκεκριμένος Γενικός Διευθυντής και η διαδικασία για την αντικατάστασή του θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η συγκεκριμένη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αγνοεί την ειδική κατάσταση της Όλαφ. Εδώ ορίζεται ο διορισμός του Διευθυντή από το άρθρο 13 του κανονισμού της ΟΛΑΦ 73 του 99 συν το άρθρο 5 της απόφασης του Συμβουλίου για την δημιουργία της ΟΛΑΦ, όπου λέγεται εκεί σε μια συναποφασισμένη ανακοίνωση ότι η διαδικασία αυτή είναι αυτή που σας περιέγραψα προηγουμένως, δεν θα την ξαναπώ. Για να διοριστεί λοιπόν ο Γενικός Διευθυντής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Αυτή είναι μια σαφέστατη απέτηση η οποία εδράζεται θα έλεγα στην κατάσταση την οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ ε, καλά σε περιπτώσεις διοργανικών υπηρεσιών όπως η ΕΠΣΟ και που δείχνει ότι η ΟΛΑΦ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Δεν είναι μια απλή γενική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διασφαλίζεται έτσι η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία της Γενικής Διεύθυνσης της ΟΛΑΦ. Όταν έχουμε να κάνουμε με την αντικατάσταση ενός τυχαίου, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, γενικού διευθυντή, σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται η λογική την οποία αναφέρει στην επιστολή της. Οπότε πρόκειται για μία παραπλευρή πρόσφορα θα λέγαμε αυτή η ανεξαρτησία και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο το διακύβημα. Η άποψή μας λοιπόν και αυτό εκφράζεται πολύ πιο ρητό στη γνωμοδότηση που πρέπει να την έχετε στα έγγραφά σας είναι πως δεν μπορούμε να παρομοιάσουμε αυτή την κατάσταση όπως κάνει η Κομισιόν σε μια φυσιολογική αντικατάσταση, σε μια φυσιολογική γενική διεύθυνση. Έχει πολύ ειδικό πλαίσιο ο Όλαφ και η ενδιάμεση αντικατάσταση χωρίς αυτό να προδικάζει το ότι η Κομισιόν πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν τη διαδικασία για να βρει έναν οριστικό αντικαταστάση σημαίνει πως πρέπει να ακολουθήσουμε το σύστημα του άρθρου 12 του κανονισμού της Όλαφ, της μουτάντης, κατά αναλογία για την ενδιάμεση αντικατάσταση δηλαδή για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία. Δεν χρειάζεται να πάμε στην επίσημη εφημερίδα αλλά πρέπει εν η Κομισιόν να ξεκινήσει μια διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να υπάρξει μια τακτική διαδικασία αντικατάστασης του κυρίου αυτού. Αυτά, σε αυτά θα ήθελα να μείνω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν ακόμα ερωτήσεις ε, προς την νομική υπηρεσία. Όχι. Οπότε το σημειώνουμε και νομίζω έχουμε στοιχεία πλέον και για τη συζήτησή μας με τον Επίτροπο. Οπότε περνάμε στο επίμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, έχουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μπονίτσι για την απαλλαγή του 2008. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μπονίτσι από το ελεγκτικό συνέδριο, τον κύριο Σεμέτα και τον κύριο Λιμπεράτσκι, τον εισηγητή μα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω τον λόγο στον κύριο Μπονίτση που έχει ετοιμάσει μια παρουσίαση PowerPoint. Yes, Thank you. Ναι, πράγματι. Κύριε Πρόεδρε, μεγάλη χαρά πάντοτε να είμαι στην Κοκομπίου που δεν ξέρω ακριβώ τι σημαίνουν τα αρχικά αυτά αλλά με μεγάλη χαρά έρχομαι. Έχω διαφάνειες να σας παρουσιάσω για την έκθεσή μου Θα περάσω λοιπόν στην πρώτη διαφάνεια. Όπως γνωρίζετε έχουμε μια γνωμοδότηση που σχετίζεται με τους λογαριασμούς που όπως ξέρετε δίνει ανεπιφύλακτη ε, γνωμοδότηση το, κοινοβου, το ελεγκτικό συνέδριο λέγοντας ότι ε, αντικατοπτρίζουν πιστά σε όλες τις ουσιαστικές πτυχές του οι λογαριασμοί, ε, οι αιτήσιοι λογαριασμοί, την οικονομική κατάσταση των κοινοτήτων από την 31η Δεκεμβρίου του 2008. Και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι δεν είναι, η πρώτη δεν είναι πάντοτε έτσι. Την πρώτη χρονιά που αντιμετωπίστηκαν ε, οι επιφυλάξεις που είχαμε στην αρχή και άρα σημειώνεται μια σημαντική πρόοδος Δεύτερον, και να μην, ε, για να μην έχουμε παρεξηγήσει. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπως ορίζονται από τη συνθήκη μόνο τη συγκεκριμένη ορολογία. Δεν σημαίνει ότι ε, δηλώνουμε μια, ε, μια αφηρημένη αξιολόγηση, αλλά το true and fair, ακριβείς και πιστές, στην ε, θετική δήλωση αξιοπιστίας είναι όρος που χρησιμοποιούμε ε, με την νομική του σημασία. Όσον αφορά τώρα την νομιμότητα και κανονικότητα. Το ελεκτικό συνέδριο γνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί προόδος και εν γέννη η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι πέρυσι Παραμένουν όμως κάποια προβληματάκια που θα αναφέρω μετά. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε ε, χρονολογική αντιπαράθεση, αντιπαραβολή και σύγκριση. Βλέπετε τα ποσοστά επί του προϋπολογισμού στον κατακόρυφο άξονα, τη ταξινόμηση με τα χρώματα κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Φυσικά το πράσινο είναι το καλό, αυτό που θα περιμέναμε, θα ήθελαμε να έχουμε το ιδεώδες. Το ποσοστό του κίτρινου ε, τμήματος, το 2,5% το ποσοστό σφάλματος έχει μειωθεί και η κίτρινη και η κόκκινη στήλη έχει επίσης μειωθεί από το 60% στο 31%. Αυτό αντικατοπτρίζει μια γενικότερη θετική εξέλιξη που θα αναπτύξω αργότερα. Χρειάζονται όμως ακόμη προσπάθειες, ιδιαίτερα όσον αφορά το κόκκινο χρώμα, δηλαδή το ποσοστό σφάλματος άνω του 5%, αλλά όχι μόνο αυτό και το κίτρινο που επίσης έχει αυξηθεί. για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με βάση τις αλλαγές που απαιτούνται. Ξέρετε βέβαια και εσείς όπως και εμείς ότι όταν υπάρχουν προβλήματα δεν υπάρχει πάντοτε μία και μόνη λύση. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Ας περάσω τώρα στον επόμενο πίνακα που έχουμε δει τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια σε δύο στήλες αυτή τη φορά. Μία που αξιολογεί τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου και πάλι βάσει παλαιότερων ετοιμάτων του Κοινοβουλίου για περισσότερες πληροφορίες ως προς την λειτουργία των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου. Και εδώ έχουμε κατανέμει σε δύο κατηγορίες. Πράσινο είναι η αποτελεσματική εποπτεία, αποτελεσματικός έλεγχος και το κίτρινο-κόκκινο είναι το κίτρινο είναι μερικώς αποτελεσματική που βλέπουμε από τα προηγούμενα χρόνια ακόμα και που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε επιπλέον προσπάθειες. Και βέβαια να κάνουμε προσπάθειες έχοντας τις υπόψη ότι δεν μπορούν να, μην, να είναι ε, μερικώς αποτελεσματικές αυτές οι δραστηριότητες ε, ιστοδύναικες. Θα πρέπει να πιέσουμε και να πείσουμε να προχωρήσουμε προς τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Έχουμε μία κόκκινη θέση, το τη συνοχή, το μη αποτελεσματικό έλεγχο, δηλαδή μη αποτελεσματική εποπτεία. Το είχαμε ήδη επισημάνει από την προηγούμενη μας ε, έκθεση, λέγαμε ότι χρειάζονται περισσότερε προσπάθειες και σημειώνω ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με, την περί... τις περιόδους 2001-2008 τα προγράμματα της περιόδους αυτά, ε, αυτής που δεν είχαν τη δυνατότητα της αντιπαραβολής και θα πρέπει σε τούτο για το μέλλον να δούμε πώς η προγραμματική περίοδος ε, που προβλέπεται από την επόμενη, στο επόμενο πακέτο μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Η Επιτροπή μας λέει, και αυτοί είναι οι διαχειριστές των προγραμμάτων, ότι έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δήλωση, γιατί πρέπει να δούμε και τα σχετικά στοιχεία. Αυτή είναι η μία πτυχή. Εν τέλει και δυστυχώς, πέρασμα αυτής της συνοχής είναι ότι δεν έχει αλλάξει η κατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια προς τη συνοχή. Για τα επόμενα χρόνια ίσως μπορούμε να περιμένουμε κάποιες καλές εξελίξεις. Ενώ άλλου τομεί που θα ήθελα να επισημάνω είναι, άλλοι τομείς που θα ήθελα να επισημάνω είναι η γεωργία που πρασίνησε. Δηλαδή μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα ε, ποσοστό σφάλματος που δεν έχει τόσο μεγάλη τόσο μεγάλε επιπτώσει, ε, δεν έχει τόσο ουσιαστικέ επιπτώσει. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για το, 15% του 5% του προπολογισμού και φυσικά κάθε σφάλμα έχει τεράστιε επιπτώσει. Και βέβαια αυτά που έχουμε διαπιστώσει σχετικά με τη γεωργία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και ω διδάγματα για τη συνοχή, για αυτά που έλεγα νωρίτερα. Ε, σε σχέση αυτά, με αυτά που μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μπρο, με αυτά που χρειάζονται να γίνουν. Καταρχάς, λοιπόν, χρειαζόμαστε καλύτερη συνολική διαχείριση και πιο αποτελεσματική χρήση των υφισταμένων πόρων εποπτείας και ελέγχου. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό και ε, πού στηρίζουμε αυτή την ε, τοποθέτηση. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για το ανεκτό ποσοστό σφάλματος, όπου αναφέρει η Επιτροπή ότι στην περίπτωση των διαρθρωτικών ταμείων το ποσοστό σφάλματος θα μπορούσε να μειωθεί σε επιπλέον, κατά επιπλέον 3% εάν χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι δομές χωρίς επιπλέον κόστος, πράγμα το οποίο εγώ προσωπικώς υποψιαζόμουν ανέκαθεν και που βέβαια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα από τους ίδιους τους διαχειριστές των προγραμμάτων ή συνδιαχειριστές για την ε, κοινή διαχείριση, Μικρή διαχείριση. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματική χρήση των υφισταμένων πόρων με, ουσιαστικές, με κάποιες βελτιώσεις, ίσως όχι ε, μεταφορά στο κίτρινο, στην κίτρινη στήλη, αλλά πάντως με καλά αποτελέσματα. Και προφανώς πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα για να βελτιώσουμε αυτή τη ε, διαχείριση σε κάθε επίπεδο και όχι μόνο να επικεντρωνόμαστε στην Επιτροπή αλλά να στραφούμε και προς το πρωτογενές επίπεδο, εκεί που γίνεται η διαχείριση του υλικού χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες εδώ. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο σε τέτοιου περιβάλλοντα να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα συνέχεια χωρίς ε, εξέλιξη. Στο δεύτερο σημείο, όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσθετου σπόρους για εποπτεία και έλεγχο με βάση μια κατάλληλη ανάλυση κόστους και αποτελέσματος. Και εδώ, Πρόεδρε, στο έγγραφο που δημοσίευσε η Επιτροπή πέρυσι, θα κάνω την παραπομπή μου, το σχετικό με, την, ε, με το αποδεκτό ποσοστό σφάλματος, όπου η Επιτροπή σημειώνει ότι το κόστος αυτό θα μπορού, των ελέγχων στην γεωργία είναι 4%, ενώ το κόστος των ελέγχων στα διαρθρωτικά ταμεία είναι κάτω του 1%. Άρα και από αυτό θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε κάποια διδάγματα. Ότι δηλαδή υπάρχει το όντι στοιχείο σχετικό με το κόστος, κοστολογικό στοιχείο ως προς την βελτίωση των ε, ελέγχων και της ε, εποπτείας. Και στα διαφορετικά σας χρειάζεται απλώς να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες. Η πρώτη μου λοιπόν πρόταση ήταν καλύτερη χρήση των υφισταμένων πόρων. Η δεύτερη μου πρόταση ήταν ότι από ό,τι φαίνεται σε όλα τα επίπεδα χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. πολλά είναι τα στοιχεία, πολλές είναι λεπτομέρειες ε, που έχουν εγγραφεί μέσα στα διαφορετικά ταμεία και αυτό συνεπάγεται περισσότερες προσπάθειες. Διαφορετικά, εμείς θα φταίμε, εμείς θα είμαστε υπέτοι εάν δεν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως και να έχουμε την καλύτερη απόδοση των χρημάτων που διαθέτουμε για τα διαφορετικά ταμεία. Αυτά σας τα λέω ως εκπρόσωπος του ελεκτικού συνεδρίου και με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχουν διαθέσει οι διαχειριστές των ταμείων. Τρίτη κατηγορία. Βελτιωσμένοι μηχανισμοί για δημοσιονομικές διορθώσεις και ανάκτηση. Στη Γεωργία βλέπουμε ότι υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι διόρθωσης των σφαλμάτων. Και μερικές φορές στρέφονται προς τον οικονομικό δικαιούχο, αλλά με, άλλε με άλλες λύσεις. Πράγμα το οποίο σημαίνει, μας περιπτώσει εν γέννη, ότι αν τυχόν διαπραχθεί ένα σφάλμα, καταβάλλεται η προσπάθεια έτσι ώστε να ανακτηθούν τα χρήματα σε οικονομικούς όρους ή μη τι άλλο να προστατευθεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν είναι οικονομικό το σφάλμα. Βλέπουμε λοιπόν κάποια πρόοδο, αλλά σημαίνω ταυτόχρονα ότι οι πληροφορίες που μας διαθέτουν τα κράτη-μέλη είναι μάλλον περιορισμένες. Υπάρχει δε μια άλλη πτυχή που θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω και είναι η έκταση των ε, επιπτώσεων, του αντίκτυπου αυτών των διορθώσεων. Να σας εξηγήσω γιατί. Εάν κάποιος κάνει ένα σφάλμα, δεν έχει καμιά επίπτωση και φυσικά δεν ε, διορθωθεί το σφάλμα, γιατί κάποιος άλλος να κάνει περισσότερες προσπάθειες. Άρα νομίζω ότι στην προσπάθεια αυτή για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων και για την ανάκτηση και πρέπει να βελτιώνει όπως έχει πράξει η Επιτροπή ήδη τις ε, πληροφορίες που διαθέτει, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και να πει ότι οι πληροφορίες που διαθέτουν τα κράτη-μέλη είναι ε, προβληματικές, είναι μάλλον περιορισμένες και άρα χρειάζεται να δούμε με πιο ξεκάθαρη ματιά το τι συμβαίνει. Είναι δύσκολο βέβαια γιατί έχουμε να κάνουμε και με, την, ε, με τα απόνερα κάποιων προγραμμάτων, με τα υπόλοιπα δηλαδή ή με μη ολοκλήρωση κάποιων προγραμμάτων όταν έπρεπε. Τώρα υπάρχουν κάποια στοιχεία απλούστευσης τα οποία βλέπουμε να εισάγονται σε ορισμένους τομείς και με καλά αποτελέσματα. Η απλούστευση λοιπόν με τα ορόσημα καταρχάς και όχι ε, με, το σύστημα των, ε, της θυμολόγησης. και έτσι μπορούμε από ό,τι φαίνεται να μειώσουμε το περιθώριο σφάλματος, απόκλησης χωρίς να περιορίζουμε το πεδίο δράση του προγράμματος, γιατί αυτό θα καταστεί αντιπαραγωγικό. Άρα έχουμε να βρούμε μια χρυσή τομή μεταξύ της απλούστευσης και της διατήρησης των λεπτομερώς περιεγραμμένων στόχων του προγράμματος. Αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για τη δική σας επιτροπή, αλλά και για τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν ανάγκη από τις λεπτομέρειες αυτές. Τέλος, όταν τα πράγματα δεν μπορούν να πληστευθούν, τότε θα πρέπει απλά να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να θεωρήσετε ε, ότι η συνέχεια του status quo δεν είναι η καλύτερη λύση. Αυτά. Grazie. Do la parola al commissario. O Kyrios Semeta, o Epitropos Semeta, è questo luogo. Mr. Chairman, rapporteur, honorable members. Provedere. Είμαι ο υπεύθυνο προτινόμενος επίτροπος για την απαλλαγή και εδώ βλέπω ότι έχω μια πολύ θετική κληρονομιά και από τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή και από το Δικαστήριο. Όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, η ετήσια έκθεση για το 2008 μας καλύπτει, δείχνοντας ότι έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες οι οποίες έχουν κακοφορήσει. Σαν αρμόδιος για τα θέματα του προϋπολογισμού, εγώ καλύπτω τα θέματα για τα οποία δεν θεωρείται απαραίτητη η ειδική τεκμηρίωση, η εξειδικευμένη τεκμηρίωση. Εδώ δεν υπάρχουν σημειωμένα σε εκκρεμότητα ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό είναι αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει. Σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο, οι λογαριασμοί περιγράφουν ακριβώς το τι έχει γίνει και τους απολογισμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια αντιμετωπίζει τα θέματα τα οποία σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχει τις προσπάθειες που κάνουν οι γενικές διευθύνσεις για να βελτιωθούν τα βασικά λογιστικά στοιχεία, βελτιώνοντας γενικότερα τις λειτουργίες της λογιστικές. Αυτά όλα περιλαμβάνονται στην προσθήκη 1. Κάτι το οποίο δεν συζητάμε πάρα πολύ συχνά, αλλά θεωρείται κρίσιμο είναι φυσικά η χρηματοδοτική πλευρά των πολιτικών μας. Το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι οι δηλώσεις των κρατών μελών και οι πληρωμές των κρατών μελών που βασίζονται στο ΑΕΠ δεν χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα λάθη, ποσοτικά λάθη. Θεωρεί επίσης ότι τα χρησιμοποιούμενα συστήματα υπολογισμού είναι γενικά ικανοποιητικά. Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει προληπτικά τις επιφυλάξεις των κρατών μελών που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα. Το κεφάλαιο 3 της έκθεσης του ελεγκτικού Συνδρίου δείχνει ότι ο βαθμός απορρόφησης των πληρωμών είναι ιδιαίτερα υψηλός, 97%. Νομίζουμε ότι αυτή η αύξηση των ποσοστών είναι ίδιον της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης οι επί του προϋπολογισμού αρχές είναι σε θέση να παρακολουθούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους, εντοπίζοντας στα πλαίσια της τρεχούσης περίοδου σε ποιους τομείς απαιτείται προσπάθεια για αύξηση των ποσοστών απορρόφησης. Οι πιστώσεις πληρωμών όμως για τη σύνοχη μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους κατά 4,5 δις λόγω της καθυστερημένης υποβολής και έγκρισης των νέων περιοδικών συστημάτων στα διάφορα Να πω επίσης ότι στο τέλος του 2009 όλα τα συστήματα αυτά έχουν γίνει δεκτά. Και έτσι και για το Ταμείο Συνοχής και για τα υπόλοιπα διαφορετικά ταμεία νομίζω ότι θα τύχουν μείωση λαθών, ποσοστού λαθών στο μέλλον. Σαν αρμόδιος για την απαλλαγή προϋπολογισμού, ε, του προϋπολογισμού γνωρίζω τις υψηλές σας προσδοκίες και φιλοδοξίες. Και αυτές ακριβώς είναι και δικές μου φιλοδοξίες και στόχοι. Θέλω να διασφαλίσω τη συνέχεια της πολύ καλής δουλειάς την οποία έκανε ο Σιμ Κάλας και όλοι οι προηγούμενοι επίτροποι Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για να το κάνω αυτό σύντομα. Καταρχάς, μείωση των περιθωρίων λάθους των ελεγκτικών συστημάτων. Δεύτερον, τα ελεγκτικά συστήματα δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν την διοικητική λειτουργία. Η πρόοδος των συγκεκριμένου αυτό τομέα θα διασφαλιστεί μέσω της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μείωση των λαθών και για τον εντοπισμό της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην απαλλαγή και στο αποδεκτό επίπεδο αν θέλετε προβλεπόμενων λαθών. Προβλεπωμένων λαθών. Δεύτερον, από κοινού διαχείριση ή προβλεπόμενων Αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί ότι έχουν υπάρξει βελτιώσεις θα έλεγα στα πλαίσια των διοικητικών λειτουργικών θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει αξία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των ελεγκτικών μηχανισμών και των ελεγκτικών δραστηριοτήτων. Θα επανεξετάσουμε τις διαδικασίες αυτές στα πλαίσια των νέων δημοσιονομικών προτινόμενων κανονισμών και θα μας ακούσετε ήδη μέσα στο 2010 περισσότερο. Σχετικά τώρα με την απλούστευση ή απλοποίηση. Πράγματι ε, τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι ιδιαίτερος περίπλοκα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια για πιο στοχευμένη χρήση. Το συνέδριο το ελεγκτικό έχει κάνει συγκεκριμένες ε, προτάσεις σχετικά με τις εφάπαξ πληρωμές, σαν παράδειγμα. Θα αξιολογήσουμε λοιπόν την επιλεξιμότητα όχι μέσω των input στοιχείων, αλλά και της απόδοσης των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Η πρώτη δυνατότητα για να κάνουμε κάτι τέτοια θα είναι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και θα προσκαλέσω τον Γιάννους Λεβαντόφσκι για να μας μεταφέρει και τις δικές του απόψεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και με τη δική σας κοινοβουλευτική επιτροπή και με τους άλλους εμπλεκομένους θα πάρω τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε τα κοινοτικά χρήματα να δαπανώνται για σωστούς λόγους και με τον σωστό τρόπο και όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους προς το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Κύριος και έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των υποχρεώσεων οι οποίες δεν έχουν ε, χρησιμοποιηθεί και μπορούν να μεταφερθούν στα επόμενα έτη στα πολιτικά προγράμματα. Αυξήθηκαν το 2008 κατά 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 12%. Ποια είναι η αποψή σας, πώς θα λυθεί αυτό το θέμα, θα, θα συνεχίσει αυτή η αύξηση των δεσμεύσεων που δεν ε, χρησιμοποιούνται, γιατί δεν είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι. Uh, thank you. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Το επίπεδο πράγματι αυξήθηκε πέρσι στα 155 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό εξηγείται γιατί αυτό είναι το ποσό περίπου δύο ετών των δαπανών δύο ετών ε, της συνοχής. Και γνωρίζουμε πως είμαστε στην αρχή ενός νέου δημοσιονομικού πλαισίου και τα κράτη-μέλη στα δύο πρώτα χρόνια ανέπτυσαν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και αυτό επηρέαζε το επίπεδο δαπανών οπότε υπήρχαν ε, υποχρεώσεις αλλά οι πληρωμές δεν ήταν τόσο γρήγορες όσο θα θέλαμε ε, και υπάρχουν ε, δύο τρόποι δύο τρόποι να μειωθεί αυτό. Ο πρώτος είναι αυτόματος. Είναι το κανόνας νη συν 2, νη συν 3 και αν ε, οι υποχρεώσεις δεν ε, χρησιμοποιηθούν εντός 2-3 ετών ε, πλέον αποδεσμεύονται, οπότε υπάρχει κάποια πειθαρχία στα κράτη-μέλη και ένας άλλος τρόπος είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία πληρωμών και εδώ πέρα καταβάλουμε πολλές ε, προσπάθειες και ε, η διαδικασία του προπολογισμού μας επιτρέπει να λάβουμε περαιτέρω μέτρα κατά τη διάρκεια του έτους. Δεν έχουμε ακόμα τελικά στοιχεία για το 2009 αλλά νομίζω πως θα δούμε ήδη κάποιες βελτιώσεις στις ε, πληρωμές ε, το 2009 και η επιτάχυνση αυτή θα μας επιτρέψει να μειώσουμε το επίπεδο των ε, αδιάθετων πιστώσεων αυτών. Σας ευχαριστώ αναφέρατε πράγματι το νήσιν 2 και νήσιν 3 δηλαδή οι δημοσιονομικές προοπτικές 1999-2006 ε, συν 3 έχει τελειώσει. 2007 συν 3 είναι το έτος στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Προσπαθήσατε να ερευνήσετε την κατάσταση με προκαταβληθέντα κονδύλια σε κράτη-μέλη. Εάν θα μπορούσαν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η κατάσταση των εσόδων του προϋπολογισμού. Ε, Μήπω χρησιμοποιήθηκαν και αυτό αντί για πραγματικές επενδύσεις. Και αν ναι, σε ποια κλίμακα έχει αυτό το φαινόμενο. As I mentioned, uh, uh, we developed, uh, όπως σας είπα χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο το οποίο ονομάζουμε έγκαιρη προειδοποίηση δημοσιονομική, budget forecast alerts. Και φυσικά κάνουμε εκθέσεις, παρουσιάσεις για τις δαπάνες αυτές και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους κάποια προγράμματα καθυστερούν στην εκτέλεσή τους. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες προμηθειών, σαν παράδειγμα, οι οποίες και αυτές δεν πηγαίνουν σχετικά γρήγορα. Η εφαρμογή κάποιων προγραμμάτων παρουσιάζει δυσλειτουργίες, χρονικά τουλάχιστον αυτό έτσι δείχνει. Και προς το τέλος του χρόνου θα έχουμε κάποια τελική ανάλυση σχετικά με το 2009. Θα την υποβάλουμε την έκθεση αυτή στις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές για να δούμε ποιες είναι καλύτερα οι αιτίε ε, για την υπό εισαγωγικά δαπάνη αυτών των πιστώσεων. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι θα κάνετε κάποιες συστάσεις προς τον κύριο Λεβαντόφσκι, ο οποίος ουσιαστικά θα σας διαδεχθεί. Τι ακριβώς έχετε στο νου σας, τι είδους προβλέψεις και συμβουλές θα δώσετε προς τον κύριο Λεβαντόφσκι για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσλειτουργίες τις οποίες αναφερθήκατε. Νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε, λέει ο κύριος Σέμετα, ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός ουσιαστικά, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, ανήκει στον αρμόδιο για τον προϋπολογισμό επίτροπο. Αυτός διαχειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ο κανονισμός ο ίδιος είναι φυσικά αντικείμενο συλλογικών αποφάσεων και το σύνολο των επιτρόπων μπορεί να κάνει προτάσεις και να συνεισφέρει και εγώ θα ήθελα να μου δοθεί δυνατότητα να κάνω κάποιες προτάσεις γιατί ασχολούμαι με τη διαχείριση του κανονισμού αυτού, του δημοσιονομικού και υπάρχουν τρία βασικά πακέτα στα οποία θα ήθελα να εμείνω. Το πρώτο πακέτο αποτελείται από την ενίσχυση του χαρακτήρα του υπολόγου θα έλεγα σχετικά με τις ευθύνες που έχουν τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στα διαρθρωτικά ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής. Το δεύτερο πακέτο αποτελείται με τις προσπάθειες και τις διαδικασίες απλούστευσης. Έχουμε πάρα πολλές ιδέες συλλέξει από τη δημόσια διαβούλευση την οποία οργανώσαμε. Από το τέλος του προηγούμενου χρόνου έχουμε ιδιαίτερα χρήσιμη γόνιμη συνεισφορά από τους εμπλεκομένους σχετικά με τις διαδικασίες απλούστευσης. Υπάρχει λοιπόν αρκετή δυνατότητα εδώ να περάσουμε σε αποτελεσματικές μορφές απλοποίησης και του δημοσιονομικού κανονισμού και των εφαρμοστικών διατάξεων και αυτά όλα θα τα μεταφέρω στον κύριο Λεβαντόφσκι. Και το τρίτο πακέτο το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει θα έλεγα να διαμορφώνεται Είναι κάποιες βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν το δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά σε αυτό το τομέα θα μου επιτρέψετε να επανέλθω σε συγκεκριμένες προτάσεις για, συ... για, τις... Ε, για τους συγκεκριμένους τομείς σχετικά με το ανώτατο αποδεκτό ποσοστό λάθους και πώς μπορεί να καθοριστεί αυτό το ποσοστό πριν κάνουμε τις προτάσεις αυτές, τις συστάσεις καλύτερα αυτές, θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε την εφαρμοσιμότητά τους βέβαια. Κύριε Επίτροπε, στις απαντήσεις που δίδεται στις γραπτές ερωτήσεις και ιδιαίτερα σχετικά με την ερώτηση παρήθμου 8 για το ανεκτό επίπεδο λάθους Είπατε ότι οι προτάσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του 2011 εκτός από την πολιτική συνοχής όπου εκεί θα υπάρξει ολοκλήρωση των προτάσεων με βάση τα στοιχεία του 2010 αλλά θα ολοκληρωθεί η διαδικασία το 2010. Το Ταμείο Συνοχής είναι ουσιαστικά το ασθενέστερο σε επίπεδο ελέγχου. Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση σχετικά με το Ταμείο Συνοχής. Και γιατί θα εμείνετε στα στοιχεία του 2010, γιατί θυμίζω ότι το 2010 καλύπτεται ουσιαστικά κατά 60% από τα προηγούμενα έτη. Και ο κανόνας αυτός, το νησιν 3, που εφαρμόστηκε για το 2007 και 2008 θα είναι ανεπαρκής για να εφαρμοστεί και το 2010. Γιατί λοιπόν αυτή η καθυστέρηση και γιατί αυτή η δυσλειτουργία. Πρώτα απ' όλα έγινε σημαντική προσπάθεια για να βελτιωθεί η νομοθεσία για τις δαπάνες της συνοχής ε, για το τρέχον ε, δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013. Και μεγάλη προσπάθεια έγινε για την εξάντε αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, εσωτερικού ελέγχου, ελεγκτικών απαιτήσεων και κανόνων στα κράτη-μέλη και θα θέλαμε να αντιληφθείτε πώς ε, τα μέτρα αυτά λειτουργούν στην πράξη και τα νομικά μέτρα. Και να αξιολογήσετε μετά την κατάσταση και το τι συνέπειες έχουν αυτά τα νομικά μέτρα για το διοικητικό κόστος και μετά να γίνουν κάποιες προτάσεις για το ανεκτό ποσοστό σφάλματος στην Κομισιόν. Για να εξηγήσω λοιπόν κάτι. Πρόσφατα κάναμε τη λεγόμενη μήνυ δήλωση αξιοπιστίας ε, στην ε, στα κονδύλια της συνοχής σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ελεγκτικού συνεδρίου και αυτή η μήνυ δήλωση αξιοπιστίας δείχνει πως ήδη έχουμε σημαντικές ε, βελτιώσεις στα συνοχή, στα της συνοχής. Προσεχώς το Φεβρουάριο δηλαδή θα σας ε, παρουσιάσουμε και κάποια έκθεση πριν τελική συζήτηση για την απαλλαγή. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Θέλουμε να υπάρξει πλήρης εφαρμογή και μετά θα φέρουμε αυτή την έννοια του ανεκτού ποστού σφάλματος στον τομέα της συνέχισης. Ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε ακόμη μία ερώτηση. Ε, θα την περιμένει βεβαίως ο κύριος Επίτροπος αφορά τον Όλαφ. Πρώτα απ' όλα, τι αναμένεται με την ημερομηνία του διορισμού νέου διευθυντή του Όλαφ ειδικά μετά τη γνωμοδότηση που ακούσαμε και ένα υποερώτημα ποιες θα είναι οι βασικές προτεραιότητες για την αναθεώρηση της νομικής βάσης του Όλαφ πώς βλέπετε εσείς να ενσωματώνετε ο Όλαφ στη δομή της Κομισιόν και σας ευχαριστώ εκ των παρτέρων Βεβαίως είμαι επίτροπος προϋπολογισμού, ακόμα δεν έχω αναλάβει τον Όλαφ. Δεν είναι ακόμα δική μου ευθύνη, αλλά όπως σας είπα λειτουργούμε συλλογικά και θα εκφράσω την άποψή μου. Πρέπει λοιπόν να γίνει διάκριση μεταξύ του διορισμού του Γενικού Διευθυντή Έχουμε πρώτα απ' όλα τον ενδιάμεσο διορισμό και μετά βεβαίως θα έχουμε και τον μόνιμο γενικό διευθυντή. Για το μόνιμο γενικό διευθυντή προετοιμάζεται η προκήρυξη της θέσης. Έχουμε ένα σχέδιο προκήρυξης ήδη και όπως ε, αναφέρω και στην επιστολή μου θα παρουσιάσουμε το σχέδιο αυτό προκήρυξης και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία. So I think uh, και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε την επιλογή και τον διορισμό νέου διευθυντή το μότερο δυνατόν. και νομίζω πως είναι κοινό μας συμφέρον να διοριστεί το στομότερο δυνατόν Γενικός Διευθυντής. Οπότε θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσω κάτι τέτοιο. Αυτό βεβαίως ε, δεν ε, εξαρτάται μόνο από την Κομισιόν αλλά από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και από το πόσο γρήγορα θα εργαστείτε. Όσον αφορά τώρα τον ενδιάμεσο Γενικό Διευθυντή, άκουσα την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, οπότε θα ήθελα να πω πως η Κομισιόν υπήρξε διάφανη σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Κάλλας απέστειλε μια επιστολή στο Κοινοβούλιο με την ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν και βλέπουμε τώρα πως και η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου διαφέρει οπότε πρέπει το συντομότερο να βρούμε μια νέα λύση για αυτό το ζήτημα και θεωρώ πως τις επόμενες μέρες θα πρέπει να συζητήσουμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό όπως ορίζει ο νόμος. Και είναι κρίμα που ο ισχύων κανονισμός δεν εξηγεί ακριβώς πώς θα αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα όταν υπάρχει ανωτέρα βία. Και πρέπει νομίζω να αλλάξει το ρυθμιστικό πλαίσιο για να προβλέψουμε και την αντικατάσταση του Γενικού Διευθυντή σε τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις. Και τέλος, για το μέλλον του Όλαφ, όπως αναφέρω και στις γραπτές μου απαντήσεις στη γραπτή μου δήλωση σκοπεύω να έχω έτοιμο ένα non-paper για το τωρινό νομοθετικό πλαίσιο γιατί νομίζω υπάρχουν κάποια επίγοντα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και σχετίζονται πρώτα απ' όλα με την ικανότητα του Όλαφ να επικοινωνεί καλύτερα με τα κράτη-μέλη στις ε, έρευνες που πρέπει να κάνει για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Όλαφ, Eurojust και Europol. Αυτό είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του Όλαφ και άλλα θέματα που νομίζω ήταν και στις καλές προτάσεις ε, του Κοινοβουλίου θα πρέπει να επανεξετάσουμε τον ισχύοντα κανονισμό για να διορθώσουμε τα εκκρεμή προβλήματα όσον αφορά τον Grazie. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουν ζητήσει τέσσερις συνάδελφοι το λόγο, όχι πάνω από 20 λεπτά, μαζί με τις απαντήσεις. Η κυρία Γιάλα Σέντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι έχω κάποιες ερωτήσεις να θέσω προς τον κύριο Μπονίτσι αλλά και προς τον ε, Επίτροπο. Η ανταλλαγή ε, πληροφοριών θα πρέπει φυσικά να αφορά και το, και το ελεγκτικό συνέδριο, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα από τα θέματα τα οποία μας ε, ενδιαφέρει αφορά και την Γενική Διεύθυνση Ρελέξ. Κύριε Μπονίτσι, για την Ρελέξ και σε επίπεδο ποσοστών ε, στους ελέγχους. Μάλλον στρέφομαι περισσότερο προς την Επιτροπή. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης των μέσων που χρησιμοποιείτε για τα RELEX. Μιλήσατε εσείς ε, όταν παρουσιάσατε τις απόψεις του ελληνικού συνεδρίου για το μέσο αγκρί. Ε, έχετε κάποιο κόστος επιπλέον να σημειώσετε για τη χρήση αυτών των νέων μέσων και ειδικά για τη ρελέξη και τις δραστηριότητές της. Το 4% των ελεγκτικών δαπανών αφιερώνεται στην γεωργία και μόνο το 1% στη συνοχή. Μήπως εκεί υπάρχει κάποια δυνατότητα βελτίωσης της ελεγκτικής παρέμβασης. Μήπως εκεί μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα το κόστος. Γιατί οι τόσο σημαντικές διαφορές στο κόστος του ελέγχου στους διάφορους μηχανισμούς και στις διάφορες πολιτικές. Για την απλούστευση την απλοποίηση μάλλον έχω ακούσει πολύ προσεκτικά το ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιλεκτικοί στα μέσα και στους στόχους ε, τους οποίους έχουμε. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να καλύψουμε ε, με διαφορετικό τρόπο κάποιους τομείς όπως ας πούμε οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες ε, είναι ο αριθμός τους πάρα πολύ μεγάλος και θα πρέπει να στοχεύσουμε σωστά. Προς τον κύριο Σεμέτα λοιπόν την Επιτροπή. Μιλάμε για την αναθεώρηση. Είπατε εσείς ότι προτιμάτε να υπάρξει σε ορισμένες περιπτώσεις μια αναθεώρηση των προγραμμάτων σχετικά με τον ανώτατο αποδεκτό κίνδυνο. Λάθος. Ε, για ποια περίοδο αναφέρετε τα στοιχεία αυτά. Ε, νομίζω ότι καλύπτουν μέχρι και το 2006. Στη συνοχή θυμάμαι ότι παλαιότερα είχε ανάψει κόκκινο φως έχει υπάρξει κάποια βελτίωση. Θα ήθελα κάπου κάπου το ελεγκτικό συνέδριο να παρουσιάζει και τις προηγούμενες περιόδους για να γνωρίζουμε τι λάθη και διορθώσεις έχουν γίνει. Επίτροπε, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γιάλο. Αναφερθήκατε σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Μου ζητάτε όμως να σας πω κάτι που δεν γνωρίζω. Το κόστος των ελέγχων δυστυχώς δεν ε, παρουσιάζεται με αρκετά λεπτομερή στοιχεία έτσι ώστε να γνωρίζουμε. Εκτός από αυτά τα οποία ανέφερα νωρίτερα για το ανεκτό ποσοστό κινδύνου όπου είδαμε πέρυσι μια έκθεση. Και αυτό που λέμε ακριβώ είναι ότι πρέπει να εξεταστεί το κόστο των ελέγχων και να εξασφαλιστεί κατάλληλη ισορροπία η χρυσή τιμή μεταξύ κόστου και αποτελέσματα. Δεν έχει νόημα να έχουμε δηλαδή πολύ ψηλό κόστο ελέγχων, να απορροφούν περισσότερου πόρου οι έλεγχοι από ό,τι τελικά κερδίζουμε με το αποτέλεσμα των ελέγχων ή κερδίζει ο πολίτη με το αποτέλεσμα των ελέγχων. Σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί η Επιτροπή σα. Και αν μου επιτρέπετε κύριε Λιπεράτη μιλήσατε για του στόχου τη συνοχή για το 2012. Όντω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, διότι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμή από τη συνοχή δείχνουν ότι το κόστο των ελέγχων κινείται σε ποσοστά κάτω του 1%. Όταν λοιπόν εδώ έχουμε και τα περισσότερα προβλήματα, τίθεται το ερώτημα, διατηρείται η ίδια κατάσταση ή μήπως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι και να βελτιώσουμε τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου. Έτσι ώστε να βελτιωθεί συνολικά η κατάσταση. Και όταν ρωτάτε γιατί να περιμένουμε στο 2012, ναι βεβαίω η ερώτηση είναι πολύ καλή. Η απάντηση από την Επιτροπή ωστόσο είναι ότι πρόκειται για νέα προγραμματική περίοδο με νέα στοιχεία που εισραίουν και βεβαίως είναι θεμητό το επιχείρημα. Πλην όμως, πλην όμως πιστεύω ότι και αν πρέπει να δώσω εγώ κάποια συμβουλή, καλό θα είναι να κοιτάξουμε τι λέει η DG Regio, η DG Employment, η την Διευθύνση για τα Περιφερειακά και την Απασχόληση και να δούμε αν οι μηχανισμοί μας επαρκούν για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αναφύονται σε 27 κράτη-μέλη. Εγώ τίνω να πω ότι μάλλον δεν επαρκούν αυτοί οι μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν αρκετοί είτε managers των διαχειριστές δηλαδή, των προγραμμάτων, είτε ελεγκτές, είτε αυτοί που θα μπορούσαν να εποπτεύουν τα προγράμματα και δεν υπάρχουν και επαρκή μέτρα πριν εμφανιστούν τα προβλήματα. Δεν λαμβάνονται αρκετά μέτρα πριν την εμφάνιση των προβλημάτων, γιατί μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλό ίσω να κάνουμε μερικά πράγματα, να εντοπίσουμε του τομεί που παρουσιάζονται τα προβλήματα, τι περισσότερε δυσκολίε και με πάντα έχοντα υπόψη την ισορροπία κόστου και αποτελέσματο, να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στου τομεί αυτού. Γιατί το όφελο θα ήταν να έχουμε περισσότερη εξοικονόμηση πόρων από του τομεί αυτού με αποτελεσματικότερα προγράμματα, με υλοποίηση των στόχων, προθέσεων, διαθέσεων του Κοινοβουλίου και ούτω καθεξής. Και άρα η αξιολόγηση αυτή βεβαίω και θα μπορούσε να περιμένει μέχρι να μα έρθουν τα πληρέστερα των στοιχείων, οι ιδεοδέστερες των συνθήκων και προποθέσεων. αλλά ίσω θα ήταν σκόπιμο να αρχίσουμε να δρούμε ήδη από τώρα, για να μην χάνουμε χρόνο. Και για την απλούστευση... Βεβαίως και δεν μπορούμε να υπεραπλουστεύουμε, δεν μπορεί δηλαδή τα χρήματα να μετατραπούν σε μια απλή δημοσιονομική μεταφορά κονδυλίων, σε ένα έμβασμα απλό. Αυτό θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα της υπερβολικής απλούστευσης. Γιατί αν κάνουμε απλώς εμβάσματα θα ε, εναπόκειται στο κράτος μέλος να διαθέσει τα χρήματα κατά το δοκούν και ίσως να μην τα βλέπει και ποτέ ο πολίτης. Άρα αυτό που υπογραμμίζει ιδιαίτερα το ελεγκτικό συνέδριο, αυτό που λέμε ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, των Ευρωπαϊκών Ταμείων σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός, ο ευρωπαϊκός, είναι διακριτός από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα προγράμματα θα πρέπει να αποβαίνουν στην βελτίωση, στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Άρα τα προγράμματα αυτά πρέπει να έχουν αυτούς τους σαφείς στόχους και όχι απλώς να είναι εμβάσματα. απλούστευση από αυτά που είπε η Επιτροπή. Βεβαίω, εγώ αισθάνθηκα μεγάλη αισιοδοξία. Πρώτη φορά είδα να ε, εκφράζεται τέτοια αποδοχή, συνένεση για τέτοιου είδου μέτρα. Μην ξεχνάτε ότι πολλοί από τους ελέγχους μας στόχο έχουν να προλάβουν την, την ε, πλευρά της εισόδου των κονδυλίων, δηλαδή να ζητούμε τα τιμολόγια, και τις προϋποθέσεις και τις περιγραφέ των δελτίων κτλ. Ενώ θα έπρεπε ίσω να κοιτάμε και την έξοδο, όχι μόνο την είσοδο των κονδυλίων, δηλαδή το πού πάνε τελικά αυτά τα λεφτά και τι ε, ε, αποτέλεσμα φέρνουν. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε ε, περισσότερη έμφαση και βλέπω ότι και η Επιτροπή δίνει κάποιε ενδείξεις που σκοπεύουν να επιφέρει αλλαγέ. Ευχαριστώ. Έχετε να προσθέσετε κάτι εσεί. Για το ερώτημα ε, που θέσατε ασφαλώς αφορά την περίοδο 94-99, την προηγούμενη περίοδο και ως εκ τούτου θα ε, πρέπει να σημειώσω ότι έχει κλείσει αυτή η προγραμματική περίοδος ήδη. Ωστόσο, πρόκειται να καταθέσουμε έκθεση για την, έκθεση, για την περίοδο αυτή. Συγκεκριμένα στις 17 Φεβρουαρίου προβλέπεται να καταθεί έκθεση. Οι προκαταρκτικές ενδείξεις όμως που έχουμε συλλέξει δείχνουν ότι το υπολοιματικό επίπεδο των σφαλμάτων στην προγραμματική αυτή περίοδο ήταν χαμηλότερο από ό,τι αναφέρεται ή ε, είχε φανεί κατά τη διάρκεια της ίδιας της προγραμματικής περίοδου. Τα τελικά όμως και οριστικά στοιχεία θα σας τα δώσουμε με την έκθεση όπως σας είπα στις 17 Φεβρουαρίου. Και αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, για να απαντήσω στον κύριο Πουνίτσα. και τις ε, ιδέες του περί ελέγχου παρακολούθησης ή καλύτερης ε, καθοδήγησης της ε, απόδοσης των δαπανών. Φυσικά και εγώ υποστηρίζω αυτή την επιλογή, να στραφούμε δηλαδή προς την ε, απόδοση, προς την έξοδο εκεί που βγαίνουν τα χρήματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου, η οποία ισχύει μέχρι πέρατος της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Άρα η εφαρμογή, η υλοποίηση τέτοιου είδους συμφωνιών, ε, σχεδίων θα πρέπει να ξεκινήσει με πιλωτικά προγράμματα πρώτα σε συγκεκριμένους τομείς για να δούμε πού ακριβώς μπορούμε να ε, εντοπίσουμε την καλύτερη περιγραφή ποια θα είναι η καλύτερη περιγραφή των, προγραμμάτων. Γιατί εάν δυσκολευόμαστε στην περιγραφή του αποτελέσματος, πώς θα ξέρουμε τι ελέγχουμε. Γι' αυτό πρέπει και να εντοπίσουμε, αυτή είναι η πρώτη δουλειά, να εντοπίσουμε τα προγράμματα με συγκεκριμένα αποτελέσματα και να τα παρακολουθήσουμε κατά τρόπο πιλωτικό ε, με μια προσέγγιση που ασφαλώς πιστεύω ότι έχει λαμπρό μέλλον μπροστά της. Σας παρακαλώ να είστε συντομότεροι γιατί θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μέρας διάταξης. Η κυρία Γκρέσλα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον καθηγητή Μπονίτσι για την αξιοπιστία των αριθμών αυτών στα γεωργικά νούμερα. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε πως 15 κράτη-μέλη έχουν κάτω από 2% αλλά 10 κράτη-μέλη πάνω από το 2% και αυτά είναι το πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε πράσινο στα αγροτικά γιατί οι άλλοι είναι τόσο καλοί. Η Γαλλία έχει 0,1, 0,2 αλλά το ανεκτό ποσοστό σφάλματος το 2% δεν σημαίνει ότι μπορούν να χαλαρώσουν αυτά τα κράτη-μέλη, γιατί πρέπει να αντισταθμίσουν τα προβληματικά κράτη και θα έρθω αυτά, όπως παραδείγματο χάρη η Ρουμανία. Ποια είναι η εμπειρία σας με τη Ρουμανία, γιατί εκεί πέρα έχουμε συστημικό πρόβλημα, έχουμε ποστό σφάλματος 12 κάτι της εκατό. Και αυτό δεν είναι καν το σωστό νούμερο, γιατί δεν υπάρχει διαχωρισμός καλλιεργήσιμης και μη γης και δεν μπορούμε καν να ορίσουμε με ακρίβεια αυτό το, το ποσοστό του σφάλματος. Οπότε θέλω να σου ρωτήσω κάτι ακόμα όσον αφορά την ανάκτηση. Ορισμένες φορές λυπούμε γιατί δεν ξέρω αν εργαζόμαστε με βάση τα τα νούμερα που, με βάση τα ίδια νούμερα που θα καταλήξουμε επίσης, να δούμε τα διευθυντικά ταμεία, έχουμε τους λογαριασμούς, στην σελίδα 82 αναφέρεται συνολικό ύψος διορθώσεων 1,277 δισεκατομμύρια ευρώ και μας είπε στο τελευταίο Στρασβούργο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής ε, πως ε, οι διορθώσεις του 2008 μόνο για τα περιφερειακά ε, ταμεία το κοινωνικό και το κοινωνικό ταμείο είναι 1,56 και έχετε εδώ πέρα για όλα τα ταμεία 1,277 και όμως μόνο για τα περιφερειακά μας είπανε 1,56 είναι 300 εκατομμύρια παραπάνω Πώς αξιόπιστη είναι αυτή η αριθμή. Εμείς σας παρακαλέσαμε μαζί με την Κομισιόν να επεξεργαστείτε ένα νέο σύστημα τουλάχιστον για την παρουσίαση των αριθμών και αυτό έγινε πριν από δύο χρόνια. Τι γίνεται ακριβώς εδώ πέρα. Να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις ανακτήσεις. Το τελευταίο κομμάτι πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί οι ε, πληροφορίες ή διαθέσιμες και η Κομισιόν κάνει αυτή την παρατήρηση πως υπάρχει κάποιος κίνδυνος αλληλεπικάλυψης μεταξύ των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη και των πληροφοριών που έχουμε και δεν είναι εύκολο να βγάλουμε τη σούμα. Οπότε το ζήτημα των ακτήσεων είναι ακόμη προβληματικό. Για να σας πω την αλήθεια, θα προτιμούσαμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα αυτές τις ε, πληροφορίες όταν ε, εξετάζουμε το ποσοστό σφάλματος, αλλά αυτό είναι δύσκολο εάν δεν είναι τόσο αξιόπιστα τα νούμερα και νομίζω ότι θέσετε το δάκλειο επί των τύπων των ήλων. Δεν μπορώ να σου ακριβώς τον λόγο, αλλά πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ αριθμών που είναι προβλέψεις, γιατί βεβαίως οι προβλέψεις τελικά δεν επαληθεύονται καμιά φορά. Οπότε αυτό είναι, αυτό είναι το, το πρόβλημα. Οπότε βελτιώθηκαν γενικά τα νούμερα στους λογαριασμούς αλλά υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις πως υπάρχει κίνδυνος άλλη επικάλυψης ε, και η, ποι... ποιότητα των δεδομένων από κάποια κρατημέλη είναι κάπως ύποπτη. Όσον αφορά τώρα τα της Γεωργίας ε, και τα κράτη-μέλη και τη Ρουμανία, εμείς δεν κάνουμε δήλωση εξοπιστίας ανά κράτος μέλος, οπότε είναι δύσκολο για εμάς να επικεντρωθούμε σε ένα κράτος μέλος. Παίρνουμε ένα τυχαίο δείγμα και δεν περιέχονται πάντα σε αυτό όλα τα κράτη-μέλη, οπότε μπορεί μερικές φορές να είναι η Ρουμανία μέσα, άλλες φορές όχι. Κατά κανόνα ε, καλύπτουμε τις, τους μεγαλύτερους ε, αυτούς παίρνουν τα περισσότερα ποσά. Ε, οπότε, εντάξει, μπορείτε να πείτε στη Γεωργία πως 15 είναι κάτω από το 2 και ίσως 10 δεν είναι, αλλά ο όγκος των ποσών είναι αντιπροσωπευτικός. Οπότε είμαστε αρκετά σίγουροι, όχι 100% αλλά λογικά στατιστικά βάσιμα ε, σίγουροι πως ε, τα νούμερα αυτά είναι σωστά για τη Ρουμανία. Αυτό το οποίο μπορώ να πω για τη Ρουμανία είναι πως αν δείτε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων των διαφόρων γενικών διευθύνσεων βλέπετε πως ε, βλέπουν προβλήματα και γίνονται εξαιρέσεις στην δήλωση αξιοπιστίας για τη Ρουμανία, καμιά φορά για τη Βουλγαρία. Οπότε φαίνεται προβληματική. Όσον αφορά τα συστήματα δηλαδή και νομίζω πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί σύν το χρόνο αναμένουμε περισσότερες πληρωμές να πάνε στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και αν τα συστήματα ήδη έχουν πρόβλημα η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Οπότε και εδώ δεν πρέπει να περιμένουμε να διωγγωθεί το πρόβλημα, πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί στη τελική ανάλυση θέμε τα χρήματα να πάνε σε αυτούς που τα χρειάζονται και να μην κόψουμε τα κονδύλια. Αλλά αυτό θα είναι ένα ακραίο μέτρο. Ελπίζω κάτι να γίνει. Να γίνει αυτή η προσπάθεια που χρειάζεται έτσι ώστε οι αρχές των χωρών αυτών να έχουν τους πόρους και τη βοήθεια που χρειάζονται για να στήσουν συστήματα τα οποία θα είναι σε θέση να απορροφήσουν αυτά τα κονδύλια. Αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Από ό,τι βλέπουμε μπορεί να είναι προβληματική η κατάσταση. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις. Ε, αν θέλετε να τις κάνετε θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ σύντομοι, συνοπτικοί και το ίδιο θα πρέπει να είναι και οι απαντήσεις οι ιδιαίτερα σύντομες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται στον καθηγητή Μποντίτσι και μετά στον Επίτροπο. Κύριε καθηγητά, το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί για το 2008 να μας πει εάν θεωρεί ότι θα έχουμε ένα τελικά θετικό δελτίο αξιοπιστίας, ε, δήλωση αξιοπιστίας ή αρνητική. Και αυτό το λέω γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πολιτικά δεδομένα. Πέρυσι είχαμε εκλογέ, είχαμε πολλές συζητήσεις, δεν θα τις ε, εκθέσω τώρα αναλυτικά, λέγαμε ότι επί 12-13 χρόνια έχουμε αρνητικό, αρνητική δήλωση. Μετά λέμε πάμε για θετική στους λογαριασμούς, αλλά για τις υποκείμενες ε, συναλλαγές δεν βλέπουμε πολύ καθαρή εικόνα και απαιτείται από τη συνθήκη μια σαφής τοποθέτηση του ελεγκτικού συνεδρίου, μια γνωμοδότηση βάσει της οποίας και εμείς ελέγχουμε την Επιτροπή και δίνουμε την απαλλαγή ή όχι. Εσείς δίνετε για τα διοικητικά, για τις διοικητικές δαπάνες ε, και την εκπαίδευση θετική δήλωση, αλλά για τη συνοχή, τη γεωργία κτλ. Δεν είναι σαφής η εικόνα. Είναι θετική ή αρνητική η δήλωση αξιοπιστίας. Και επίσης, για τον Επίτροπο Σεμέτα, τον οποίο καλωσορίζω εδώ, είπατε ότι βελτιώνονται, βελτιώνονται χάρη στο ελεκτικό συνέδριο και του συναδέλφου σα, ε, οι λογαριασμοί είναι βεβαίω, αλλά χάρη στην Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού επίση. Γιατί αν δείτε τα τελευταία χρόνια τι είδου πιέσει ασκούν στην Επιτροπή σα, στην Εκτελεστική Επιτροπή, οι βουλευτέ και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, ασφαλώ θα συμφωνήσετε ότι είναι στην πηγή αυτών των βελτιώσεων οι ευρωβουλευτέ. Και επίση, είχατε μιλήσει για τον στόχο μιας θετικής δήλωσης αξιοπιστίας. Έχουμε τη συνήθεια ο πρόεδρος της Επιτροπής να μας υπόσχεται μια θετική δήλωση αξιοπιστίας. Το ίδιο είναι, χωρίς επιφύλαξη ή θετική, το σημειώνω αυτό. Και βλέπουμε η κοινή γνώμη να τίνει προς μια κατάσταση κατά την οποία φαίνεται ότι δεν ελέγχεται η ε, ο δημόσιος τομέας, το δημόσιο. Ο δημόσιος έλεγχος δηλαδή δεν είναι ικανοποιητικός. Και βλέπουμε μερικές φορές θετικές δηλώσεις αξιοπιστίας, αλλά με επιφυλάξεις. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, εάν τα καταφέρνουμε τόσο το καλύτερο. Ή αλλιώ αν έχω μια μικρό δήλωση αξιοπιστία, mini DAS. Και ίσω τότε να έχετε πρόβλημα ε, ανεξαρτησίας εσείς. Αν αναπτυχθεί αυτή η έννοια της μήνυ δήλωση αξιοπιστίας, που ίσως δεν είναι κακή ιδέα, θα έχουμε έναν τρόπο να διατηρήσουμε τον έλεγχο μέσω του ελεκτικού συνεδρίου με τους διαρκείς ελέγχους. Δεν ήταν σύντομη η ερώτησή σας, λέει ο Πρόεδρος. Όπως και ο κ. Κοτσολίνο θα πρέπει να φύγει πάρα πολύ σύντομα. Θα απαντήσει ε, πολύ γρήγορα ο Επίτροπος Σεμέτα και ο εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να παραμείνει μετά ε, ο κύριος Επίτροπος για να δώσει και τις δύο άλλες ε, απαντήσεις. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος λοιπόν. Είναι σαφές ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να μην θέτουμε στόχους τους οποίους δεν μπορούμε να πετύχουμε. Πρέπει να βάζουμε πάντα στόχους τους οποίους, προς τους οποίους μπορούμε να κινηθούμε έτσι ώστε να πετύχουμε όσο περισσότερα πολλά μπορούμε και οι θετικές δάσεις, οι θετικές δηλώσεις αξιοπιστίας πρέπει να είναι βασικός στόχος από εδώ και πέρα. Οι δηλώσεις αξιοπιστίας για να είναι όλες θετικές ε, νομίζω ότι είναι ένας πολύ ε, φιλόδοξος στόχος αλλά έχει σημειωθεί πρόοδος μπορώ να είμαι αισιόδοξο. Ο κύριος Μπονίτσι. Η απάντηση είναι περίπλοκη. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά α, πρέπει να πω ότι εδώ και 12 χρόνια το ελεγκτικό συνέδριο έπαιρνε ένα υπόδειγμα από το σύνολο του προϋπολογισμού και τότε μπορούσε κανείς να μιλήσει πολύ εύκολα για μια θετική ή μια αρνητική δήλωση. Από τότε όμως έχουμε περάσει σε διαδικασίες αποσπασματοποίησης των σημείων ελέγχου στον προϋπολογισμό και έχουμε πολλαπλές γνωμοδοτήσεις που αφορούν τη γεωργία, που αφορούν ε, τη συνοχή και το να αναφέρει κανείς ε, μία και μόνο φράση, θετική ή αρνητική, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα ήθελα να προτείνω ότι θα πρέπει να μιλάμε και για τις αποχρώσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στις απαντήσεις οι οποίες δίδονται. Θα πρέπει επίσης να αναφερόμεθα και στις αλλαγές οι οποίες έχουν επισυμβεί γιατί τώρα πια έχουμε μια εικόνα κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου χρόνου θα έλεγα, μιας μεγάλης χρονικής περίοδου. Και δεν μπορούμε να δώσουμε μια μονολεκτική απάντηση. Όταν ξεκίνησα την πρώτη μου εντολή πριν έξι χρόνια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να έχει ένα πράσινο φως στη Γεωργία. Τώρα το έχουμε το πράσινο φως στη Γεωργία. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι εξελίσεις και ποιες οι αποχρώσεις και τι πρόοδος έχει τελικά συντελεστεί. Δεν νομίζω ότι από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να αλλάξει το φως αυτό, το χρώμα αυτό. Πράγματι πριν πέντε χρόνια μπορεί να υπήρχε μία κάπως πιο μονολεκτική σε εισαγωγικά απάντηση, αλλά τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Και αυτή είναι και η τάση στους διεθνείς ελεκτικούς μηχανισμούς να κοιτάει κανείς την εξέλιξη των πραγμάτων και να μην βλέπει σαν να δικαστεί σε μπάση περιπτώσει τα πράγματα για να πει στο τέλος ναι ή όχι, ένοχος ή αθώος. Καλώς. Όπως είπα ο κύριος Κοτσολίνος ζήτησε την δυνατότητα να μιλήσει νωρίτερα και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο Σεμέτα να μείνει στην αίθουσα για να δώσει απαντήσεις στους δύο βουλευτές οι οποίοι ακόμα δεν έχουν προλάβει να τις Ο κύριος Κοτσολίνο θα μας μιλήσει για το θέμα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων. Και καλωσορίζω και τον Επίτροπο κύριο Κάλλας. Σας ζητώ συγγνώμη, λέει ο κύριος Κοτσολίνο, αλλά επικαλύπτονται κάποιες ε, εργασίες τις οποίες πρέπει να κάνω και γι' αυτό ζήτησα να μιλήσω νωρίτερα. Το ένα το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι η ευαισθητοποίηση των κρατών μελών σε σχέση με την πρόληψη των απατών και των μη κανονικών διαδικασιών, των παρατυπιών. Και επίσης να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να καταστήσουμε τους ίδιους πόρους πιο αποτελεσματικούς σε σχέση με τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε είτε στο εσωτερικό της Ένωσης είτε στο εξωτερικό. Γι' αυτό ακριβώς η έκθεση την οποία παρουσιάζω λαμβάνει υπόψη τις ε, συζητήσεις που έγιναν με την ΟΛΑΦ, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις συναντήσεις με τον Σκιώδη Συγητή, με τον οποίο θα έλεγα έχουμε σαν βασικό στόχο και οι δύο το να καταστήσουμε πιο διαφανείς τις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών. Σημειώνουμε μία τάση σε όλους τους τομείς Μία βελτίωση σε σχέση με τις εκτιμόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις από τις παρατυπίες και από τις απάτες. Έχει υπάρξει βελτίωση και περισσότερο έχουμε να κάνουμε με λάθη και όχι τόσο με υποψίες απατών και αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς και για όλα τα κράτη-μέλη. Σε σχέση με τους ιδίους πόρους θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των στατιστικών στοιχείων τα οποία παρέχουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Το θέμα της διοικητικής συνεργασίας στον φορολογικό τομέα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Η πρόταση του Συμβουλίου είναι ένα πρώτο βήμα. Παραμένει η ανάγκη να ελέγξουμε καλύτερα τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ίδια τα κράτη-μέλη δεν συνεργάζονται και να δούμε επίσης και ποιο είναι το κόστος των συμπληρωματικών μέτρων για τους ιδίους πόρους στα διάφορα κράτη-μέλη και τι αντισταθμίσεις μπορεί να υπάρξουν. Για τις γεωργικές δαπάνες έχει υπάρξει μία μείωση των παρατυπιών κατά 34% σε σχέση από το 2007. Πρόκειται για μία μείωση των απατών η οποία οφείλεται ταυτόχρονα και στον υψηλότερο αριθμό των περιπτώσεων οι οποίες καταγγέλθηκαν και εξετάστηκαν. Θα πρέπει εμείς να καταστήσουμε πιο ε, αυστηρή την εκτέλεση του κοινωνικού κανονισμού ε, Κατά 27% ε, σημειώνονται λιγότερες ε, παρατυπίες και λάθη και για τα διαρθρωτικά μέτρα και τα διαρθρωτικά ταμεία. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια σε εισαγωγικά αυστηροποίηση των τρόπων σεβασμού και των μεθόδων σεβασμού του κανονισμού, όπως το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο. Θα πρέπει να υπάρξει μια σωστότερη επίσης μορφή ε, ελέγχου των ποσοτικών στόχων τους οποίους έχουμε θέσει χωρίς να αγνοούμε την ποιότητα γιατί πολλές φορές εμένουμε σε ποσοτικά στοιχεία και αγνοούμε την ουσία. Διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχει μία μη ομοιογενής ε, διάθεση συνεργασίας από τα κράτη-μέλη. Έχουμε πολύ ελλειπτικές πληροφορίες σχετικά επίσης για την περίοδο 2000 με 2006. Η συγκεκριμένη στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των απατών σε συνεργασία με την ΟΛΑΦ είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Πάντα μιλάω για τα διαρθρωτικά ταμεία. Σχετικά με τα προενταξιακά ταμεία έχουμε κάποια προβλήματα πιο σοβαρά βέβαια θα πρέπει να ενισχύσουμε την διοικητική ικανότητα των συγκεκριμένων χωρών να διαχειριστούν τα κοινοτικά χρήματα, τις κοινοτικές πιστώσεις. Θα πρέπει να αποφύγουμε συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των συγκεκριμένων πιστώσεων και σε εθνικό και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Για τις άμεσες δαπάνες έχουμε πολλά προβλήματα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της διπλής χρηματοδότησης ορισμένων προγραμμάτων για διοικητικούς λόγους. Έχουν γίνει κάποια βήματα για ένα ελεγκτικό πλαίσιο εσωτερικό πιο ολοκληρωμένο ιδιαίτερα σχετικά με το ανεκτό ποσοστό ε, λάθος. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των στοιχείων που δίδουν στα κράτη-μέλη να έχουν μια πιο σταθερή νομική βάση και να παρουσιάζουν όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά το αποτέλεσμα των ελεγκτικών ενεργειών που διατάσσονται στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Και εδώ η κατάσταση της ΟΛΑΦ φυσικά έχει άμεσο ρόλο με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων ε, χρειάζεται καλύτερη επάνδρωση της ΟΛΑΦ έτσι ώστε διοικητικά να λειτουργεί πιο άνετα. Ε, πρέπει να είναι η έλεγχη πιο αποτελεσματική από ό,τι σήμερα και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια κατελάχιστον κοινή πολιτική η οποία θα επιτρέψει τη σύγκριση των στοιχείων και θα επιτρέψει επίσης και τη συνεργασία ανάμεσα στην ΟΛΑΦ και τις εθνικές ελεγκτικές αλλά και δικαστικές αρχές. Το θέμα της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές παραμένει ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα και γι' αυτό ακριβώς θα μας επιτρέψετε να προτείνουμε και μέσω των τροπολογιών οι οποίες έχουν κατατεθεί για την ΟΛΑΦ να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να υπάρξουν ε, έλεγχοι στις στρατηγικές οι οποίες ακολουθούνται στα διάφορα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των παρατυπιών και των απατών. Είναι μια ανάλυση η οποία φαίνεται απαραίτητη για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα η ΟΛΑΦ και κυρίως να μπορέσουν οι έλεγχοι να γίνουν με πιο συμβατό μεταξύ τους τρόπο σε όλες τις χώρες θα είναι και το πρώτο βήμα για τον καθορισμό μιας πραγματικής προσπάθειας ορισμού των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια της προστασίας των συμφερόντων αυτών. Αν θέλουμε πράγματι να συνεισφέρουμε με αποτελεσματικό τρόπο στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανονισμών, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε τα στοιχεία τα οποία μας θέτουν στη διάθεσή μας ε, οι διάφορες χώρες μέλη, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να διαμορφώνουμε σε κοινοτικό επίπεδο τις πολιτικές, ε, ε, ιδιαίτερα τις πολιτικές συνοχές. Οι πολιτικές συνοχές υποφέρουν θα έλεγα και στο σχεδιασμό τους και στη φάση σχεδιασμού από τις τρευλώσεις τις οποίες οδηγούν τα στοιχεία και ο τρόπος συλλογής των στοιχείων αυτών. Ευχαριστώ κύριε Κοτσολίνο, μας τα παρουσιάσατε όλα πάρα πολύ συνοπτικά και συνθετικά. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση για την έκθεση Κοτσολίνο, επιστρέφουμε στην ε, έκθεση σε μέτα και ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Αντρέασεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα μια ερώτηση για τον κύριο Πονίτσι. Είπατε πως όταν λέμε unfair μπορούμε αυτό να το αντικαταστήσουμε με το fair το οποίο δεν ισχύει Ισχύει ότι αυτό έγινε στου ελευθερού λογαριασμού και θα μπορούσατε να το κάνετε όταν λέτε στην παράγραφο 8 πως υπάρχουν αδυναμίες στο λογιστικό σύστημα που θέτουν να αμφιβόλω την ποιότητα των πληροφοριών σε κάποιες γενικές διευθύνσεις. Προς τον κύριο Σεμέτα τώρα. Απαντώντας ε, στην αξιοπιστία μιλήσατε για κάποια επιτεύγματα και μιλήσατε για ένα δίκτυο λογιστικής, ε, λογιστικών ανταποκριτών. Είναι επίτευγμα αυτό, είναι ένα βήμα στην όλη διαδικασία επίδομα θα ήταν η βελτίωση της ποιότητας ε, των πληροφοριών. Όσον αφορά... Στην ίδια απάντηση λέτε πως ε, ο επικεφαλής ε, λογιστής δεν επικύρωσε τα συστήματα τα λογιστικά της Ρέλεξ. Χτες ή προχτές ακούσαμε τον αρμόδιο και μας είπαν οι ελεγκτές πως υπάρχουν πάρα πολλά σφάλματα εκεί πέρα. Πώς είναι δυνατόν μετά από 10 χρόνια από την διοικητική μεταρρύθμιση δεν έχει γίνει τίποτα για να βελτιωθούν τα συστήματα της Relax. Όσον αφορά τις προτεραιότητες για το ανεκτό ποσοστό σφάλματος έχουμε πάει από την μηδενική ανοχή του πρώτη σε ανεκτό επίπεδο σφάλματος. Νομίζω πως εδώ πέρα μειώνεται το επίπεδο των διαβεβαιώσεων που δίνουμε στους φορολογούμενους. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συνέβη αυτό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Έχει κλείσει η συζήτηση για την έκθεση που συζητάμε τώρα και δεν θα γίνει σωστή συζήτηση για την έκθεση Κοτσολίνο. Ο εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου Μπονί. Θα είμαι πολύ στόμο. Έχουμε θετική δήλωση αξιοπιστία χωρί επιφυλάξεις και χωρίς ε, ιδιαίτερη υπόδειξη που είχαμε στο παρελθόν σημειώσει. Και πρέπει να σημειώσω ότι στο ελεγκτικό συνέδριο, όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό, υπό τη δική μου Προεδρία, είχαμε την επιλογή να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία true and fair, τους όρους true and fair, ή αυτή την ορολογία που χρησιμοποιήσαμε εδώ. Αλλά Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς την χρήση των όρων αυτών. Του χρόνου τι θα κάνουμε δεν ξέρω να σας προβλέψω. Θα πρέπει να ρωτήσετε εκείνον που θα έχει αναλάβει τον τομέα αυτό όταν έρθει η στιγμή. Σας ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Σεμέτα. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος. Ως προς την αντιστοιχία των λογαριασμών. Βλέπουμε αυτή την εξέλιξη ως πολύ, θετική εξέλιξη. Επεκτείνεται διαρκώς η αντιστοιχεία. οι ανταποκριτέ ε, για του λογαριασμού και αυτό βέβαια μα επιτρέπει με ένα καλύτερο δίκτυο να βελτιώσουμε και την ε, ε, νοοτροπία τη σχετική με την τήρηση των λογαριασμών στην Επιτροπή. Θα ήθελα να σημειώσω ότι πάνω απ' όλα ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας, μια νέα προσέγγιση την οποία φυσικά θα πρέπει να προαγάγουμε ενισχύοντας και συνεχίζοντας την εκπαίδευση, την κατάρτιση για τους λογιστές μας και, τα... και χάρη σε αυτό το λογιστικό δίκτυο ή δίκτυο λογιστών. Ως προς τη ρέλεξη μπορώ να πω ότι το όντι ο επικεφαλής του λογιστικού γραφείου δεν ενέκρινε, δεν έδωσε τελική ε, πιστοποίηση στους λογαριασμούς της Ρέλεξ, πλην όμως υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στους τομείς αυτών των λογαριασμών, πλην ορισμένων όπου χρειάζεται ακόμη περισσότερη βελτίωση, αλλά πάντως είμαστε κάτω από το επίπεδο του ουσιαστικού σφάλματος. Και πιστεύω ότι στο μέλλον θα μπορούμε να κυρώνουμε και τα, τα συστήματα λογαριασμών του οικογένειας Ρέλεξ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με βάση τα δεδομένα του τομέα της ενέργειας και των μεταφορών βλέπουμε ότι έχουμε ένα ποσοστό σφάλματος ε, ύψους 5%. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η αναθεώρηση των πολύ περίπλοκων όντως ε, διαδικασιών που αφορούν και την ε, κατανομή αλλά και την απορρόφηση των κονδυλίων. Και επίσης άλλη μια ερώτηση ως προς τις αντικανονικές και παράνομες ε, συναλλαγές. Πιστεύω ότι αυτές θα έπρεπε να καταγγέλλονται στο δημόσιο χώρο πολύ περισσότερο. Θα πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει που τα κονδύλια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει. Δυστυχώς όμως σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένα ε, κοινά θα έλεγα, ομάδες της κοινή γνώμης σε ορισμένες χώρες δεν φτάνουν αυτές οι πληροφορίες. Άρα καλό θα ήταν και στην αρχή του έτους να δημοσιοποιούνται αυτά τα προβλήματα με την ελπίδα ότι θα έχουν παραδειγματικό αποτέλεσμα ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον τα σφάλματα. Και πιστεύω ότι και το κοινό θα βοηθούσε με τη συμπεριφορά του στην αποφυγή των σφαλμάτων προ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μπορώ να είμαι σύντομο για την ενέργεια και τι μεταφορέ. Έχουμε ένα ποσοστό σφάλματο 2-5%. Κάπου εκεί βρισκόμαστε. Ε, δεν είναι απαραίτητα στο υψηλότερο επίπεδο, το 5% δηλαδή το σφάλμα, μπορεί να είναι και κάπου στη μέση προ τα κάτω. Και πάντω είναι ένα τομέα αυτό τη ενέργεια και των μεταφορών που έχει σημειώσει βελτίωση, με, έχει χαμηλότερο ποσοστό σφάλματο από ό,τι στο παρελθόν, χωρί βέβαια να έχει επιτύχει το ποσοστό που θα ήταν κάτω του 2%, δηλαδή που θα επέτρεπε να το χρωματίσουμε πράσινο. Και πάλι στον τομέα αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσαμε πολλά να κερδίσουμε χάρη στην απλούστευση. Γιατί είναι αρκετοί οι κανονισμοί στον τομέα αυτών που είναι περίπλοκοι. Κύριο Σέματα, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος για την ενέργεια και τις μεταφορές νομίζω βλέποντας την ε, απλώστευση, την απλούστευση όπως προτείνεται και προβάλλεται δεν σχετίζεται μόνο με την πολιτική συνοχή ή το, τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και τις μεταφορές, την ενέργεια που θα αγγίξει η απλούστευση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο δημοσιονομικός κανονισμό έχει εγκάρσια ε, διατύπωση. Φυσικά για συγκεκριμένους τύπους νομοθεσίας απαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την τροποποίηση των κανονισμών, παραδείγματι υπάρχουν σε άλλα σημεία περισσότερο, πιο εύκολες διατάξεις, πιο απλές διατάξεις ε, από ό,τι τροποποίησεις στο δημοσιονομικό κανονισμό ή Ε, αλλά πάντως κάθε βελτίωση στον δημοσιονομικό κανονισμό θα σημάνει ε, εφαρμογή και στους ε, λοιπούς εμπλεκόμενους τομείς. Ω προ την καταγγελία στην κοινή γνώμη, θα συμφωνήσω μέσα ότι η διαφάνεια θα μα βοηθήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή το σύστημα της ε, δημόσιας κατακραυγής, δηλαδή καταγράφουν οι γενικοί διευθυντές μας στο τέλος του χρόνου τα κράτη τα οποία δεν έχουν ε, ε, τηρήσει τις προϋποθέσεις των κανονισμών και βέβαια και στην έκθεση για το 2008 είχαμε προεξαγγείλει τα κράτη-μέλη τα οποία δεν πληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις. Συμφωνώ μας μαζί σας ότι θα μπορούσαμε να περιμένουμε να εξασφαλίσουμε και περισσότερη πρόοδο. Κυρία Γκρέσλε, για 30 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω στον κύριο Σέμετα πως πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, σοβαρά την ε, απάντηση της νομικής υπηρεσίας. Κάθε μέρα που περνάει κινδυνεύει η νομιμότητα του Γενικού Διευθυντή του Όλαφ. Και κανείς δεν θα ρωτήσει τότε εάν ήσασταν ή δεν ήσασταν ακόμα επισήμως επιτρόπος. Οπότε θέλω επιγόντως μία απάντηση. Ευχαριστώ κύριος Κάλλας για την έκθεση Κοτσολίνο και ευχαριστούμε τον κύριο Σεμέτα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ λοιπόν και τον εισηγητή. Ευχαριστώ επίσης και για την επιμονή σας στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ γιατί κρατήσατε πολύ ψηλά στις προτεραιότητές σας και την καταπολέμηση των απατών και παρατυπιών. Σας ευχαριστώ και για την έκθεσή σας, η οποία παίρνει στοιχεία από τις εκθέσεις της ΟΛΑΦ. Και προσπαθούμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τη διαχείριση των κοινοτικών χρημάτων και θα συνεχίσουμε επίσης και την διαμόρφωση του εσωτερικού πλαισίου ελέγχου στους κεντρικούς πολιτικούς τομείς, στους κεντρικούς τομείς πολιτικής μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν, όπως και οι μορφές συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, για να γίνει η σχέση ανάμεσα στις δικαιτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες αποτελεσματικότερη και χρησιμότερη και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το ελεγκτικό αυτό πλαίσιο. Βλέπουμε στην έκθεσή σας ότι αναγνωρίζεται η μακρόχρονη συνεργασία ανάμεσα στην ΟΛΑΦ και τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίδονται παραδείγματα στα διαφορετικά ταμεία και στην εξωτερική βοήθεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα μας βοηθά ζητώντας από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους έχει υπάρξει σαφής, αργή αλλά σαφής βελτίωση στα πλαίσια της συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, στα πλαίσια της πρακτικής name and shame, δημόσιας καταγγελίας δηλαδή, έχει υπάρξει κάποια πρόοδος και αυτό έχει θετικά αποτελέσματα και στην προστασία των ε, οικονομικών συμφερόντων. Το άρθρο 325 ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις ενέργειές τους για να προστατεύσουν τον δημοσιονομικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα κατανομής αρμοδιοτήτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρατη από κοινού προσπαθούν να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα αυτά. Η έκθεση παρουσιάζει ιδιαίτερα κάποιες στατιστικές σε σχέση με απάτες και παρατυπίες. Οι στατιστικές αυτές οι οποίες παρουσιάζονται στο, σύμφωνα με το άρθρο 325 βασίζονται στις εκθέσεις τις οποίες μεταφέρουν τα κράτη-μέλη. Καλύπτουν όλους τους τομείς ε, του κοινοτικού προϋπολογισμού. Παρουσιάζει η έκθεση αυτή και στατιστικές για τις δαπάνες οι οποίες ελέγχονται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι στατιστικές αυτές, τα στατιστικά αυτά στοιχεία ε, είναι άμεσο ενδιαφέροντος για το κοινό και για τον τύπο και είναι θα έλεγα η έκθεση αυτή μία από τις λίγες πηγές οι οποίες δίδουν στοιχεία σχετικά με την καταπολέμηση των δαπανών και των παρατυπιών. Θα πρέπει όμως να γίνουν αντικείμενο προσεκτικής διαχείρισης και αντιμετώπισης αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παρατυπιών ε, και όχι θελημένων απατών βέβαια, όπου εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά και μια απάτη δεν χαρακτηρίζεται σαν τέτοια παρά μόνο εφόσον υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Οι οικονομικές επιπτώσεις των απανών μπορούν να προσμετρηθούν μόνο στο τέλος των δικαστικών διαδικασιών. Ξέρω ότι τα θέματα αυτά συζητιόνται κάθε φορά και κάθε χρόνο όταν συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά εμείς προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να καταστήσουμε το πλαίσιο πιο ευκρινές γιατί παραμένει ιδιαίτερα περίπλοκο. Ευχαριστώ. Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είμαι αναπληρωτής και σκιώδης ηγητής στην έκθεση Κοτσολίνο και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την έκθεσή του και για τα σχόλια του Επιτρόπου. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με τα σχόλια που άκουσα από την κυρία Ανδρέασεν. Καμιά φορά νομίζω είναι πολύ καλό αυτό το οποίο κάνετε που ασχείτε κριτική στους πάντες συνέχεια. Χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Αλλά δεν θα μπορούσατε όταν υπάρχουν θετικές εξελίξεις, όταν υπάρχουν βελτιώσεις, δεν θα μπορούσατε να το αναφέρετε. Δεν θα είναι έτσι λίγο και πιο αξιόπιστη κριτική σας. Διαβάζω τα βιβλία σας, μελετώ τα ποια έχετε κάνει. Ε, χρειαζόμαστε συναδέλφους σαν και εσάς, αλλά καμία φορά μπορείτε να πείτε τουλάχιστον πως είναι μισογεμάτο καμιά φορά το, το ποτήρι και όχι μόνο ε, μισοάδιο. Βεβαίως η απάτη είναι πολύ σοβαρή, ειδικά όταν μιλάμε για δημόσια κονδύλια Οπότε παίζουν σημαντικό ρόλο και οι ελεγκτές και οι διαχειριστές για να καταπολεμηθεί να καταπολεμηθούν οι παρατυπίες. Οποιαδήποτε κατάχρηση των γενετικών κονδυλίων είναι απαράδεκτη και βέβαια πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή. Πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για περαιτέρω διαφάνεια εντός της Ένωσης και το αναφέρεται και αυτό. Ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ακριβώς η αναγνώριση των συνεισφορών πως όπως παραδείγματο χάρη οι αγροτικές επιδοτήσεις πρέπει να είναι διαφανής μέχρι το τελευταίο ευρώ. Επίσης πρέπει να σφίξουν τα λουριά όσον αφορά την διαχείριση από τα κράτη-μέλη καθώς οποιοδήποτε ευρώ ε, χρησιμοποιείται άδικα ή οποιαδήποτε κορώνα μια που είμαι Σουηδός έχει κλαπεί από το φορολογούμενο πρέπει να αξιολογήσουμε καλύτερα τον κίνδυνο να δράσουμε κατά της απάτης στην παραμικρή υποψία παρατυπίας να επικεντρωθούμε στις ε, διαρθρωτικές βελτιώσεις που χρειάζονται για παρακολούθηση των παρατυπιών και νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αν δεν λέει κανεί καλά λόγια στον Επίτροπο θα τα πω εγώ. Νομίζω πως ήταν πολύ καλός ο Επίτροπος. τουλάχιστον αν δείτε από πού ξεκίνησε. Αυτό επιτυχάνεται μέσω σαφών προτεραιοτήτων και μπορούμε να το πούμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, ούτε και η χώρα μου έχει κάποια προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να φέρουμε αυτά τα προβλήματα στην επιφάνεια, να τα συζητήσουμε και να διορθώσουμε τα λάθη. Και εδώ, κυρία Ανδρέασεν, έρχεστε εσείς να μην επαναλαμβάνονται συνεχώς οι ίδιες υποθέσεις και έχουμε δει βελτιώσεις. Κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Σημαντικό είναι να δούμε τις πληροφορίες της έκθεσης για τα προενταξιακά κονδύλια. Στη χώρα μου, στο Σουηδικό ραδιόφωνο, πριν από λίγες εβδομάδες, κάποιοι δημοσιογράφοι έλεγαν πως η προενταξιακή βοήθεια για την Τουρκία είχε πάρα πολλά κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν λάθος, δεν πάνε σωστά μέρη, δεν δίνονται σε μειονότητες. Ίσως αυτό να είναι πρόβλημα κυρίως Τουρκίας θα έλεγα ότι είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στον τομέα αυτό, μαζί με, τους, ε, μαζί με τον σοσιαλδημοκράτη συναδελφό μου, τον κύριο Γιώργο Φάν, στείλαμε μια επιστολή στον κύριο Λιρέν και ελπίζω τις τελευταίες ημέρες που έχει το αξίωμά του να στείλει μια επιστολή και ελπίζω να λάβετε και σε ένα αντιγραφή κύριε Κάλλας. Η υποχρέωση δημοσίευσης ε, το πώς, του πώς διανέμονται τα κονδύλια. Πρέπει να διευρυνθεί και να ισχύει για όλα τα κρατη που έχουν λάβει στήριξη. Και πρέπει επίσης να νομοθετήσουμε την δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας και στο δημόσιο τομέα. Τέλος, ε, κύριε Εισηγήτα και κύριε Επίτροπε, στην έκθεσή σας στο σημείο 5.2, έκθεση για τη Γεωργία, σελίδα 27, αναφέρεται το μηχανισμό, τον αυτόματο μηχανισμό εκαθάρισης στο άρθρο 32 του κανονισμού του Συμβουλίου. Μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί με πιο αυστηρό τρόπο, γιατί νομίζω πως οι φορολογούμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη ίσως μπορούν να συμβιβαστούν με το ότι υπάρχουν προβλήματα με κάποια από αυτά τα ταμεία, ειδικά σε κάποιες χώρες, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να αποδεχτούν μακροπρόθεσμα ότι δεν κάνουμε αρκετά για να ανακτήσουμε τα κονδύλια. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή και να ρωτήσω τον, τον Επιτροπό εάν το άρθρο αυτό και το σύστημα μπορεί να ερμηνευθεί και να χρησιμοποιηθεί αυστηρότερα. Ευχαριστώ και νομίζω έχετε κάνει καλή δουλειά κύριε η συγητά. Η κυρία Γκρέσλε. Και εγώ λέει η κυρία Μακοβέη αντί για την κυρία Γκρέσλε ότι η έκθεση αυτή είναι μια καλή έκθεση και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπορέσαμε να συνεργαστούμε επανειλημμένα με τον κύριο Κοτσολίνο στα πλαίσια της έκθεσής του. Αυτό το οποίο έχει σημασία να αναφέρουμε εδώ είναι οι δημόσιες προμήθειες. Είναι ένας από τους τομείς ο οποίος είναι ο πιο ευάλωτος θα έλεγα για κακή διαχείριση και για περιπτώσεις διαφθοράς. θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για τις δημόσιες προμήθειες. Στα πλαίσια του τομέα πάντα των δημοσίων προμηθειών θα πρέπει να δούμε τι εθνικά μέτρα λαμβάνονται για να διασφαλιστεί το υπόλογο και η διαφάνεια και θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε σε εθνικό επίπεδο τα ελεγκτικά συστήματα πάντα σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες. Για να προλάβουμε τις απάτες αυτό που έχει σημασία είναι η διαφάνεια. Οι δικαιούχοι των Ευρωπαϊκών Ταμείων θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι πάντα να δίδουν όλες τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται. Το 20% του κοινοτικού προϋπολογισμού περνάει φυσικά από τα διαρθρωτικά ταμεία, ενώ το 80% το οποίο πολλές φορές δίδεται είτε από τον υπόλοιπο κοινοτικό προϋπολογισμό είτε από τους εθνικούς προϋπολογισμούς δεν οφείλει να δίδει τα στοιχεία τα οποία οφείλει να δίδει το 20%. Θα πρέπει αυτός, αυτή η νομική ρύθμιση να βελτιωθεί έτσι ώστε όλοι οι δικαιούχοι να είναι γνωστοί σε μία ιστοσελίδα σαν παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει τα στοιχεία τα οποία δίδουν τα κράτη-μέλη, τα οποία θα ενημερώνουν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα να είναι υπεύθυνα και σωστά. Ζητάμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου το σύστημα από κοινού διαχείρισης και να μας κάνει μια έκθεση γύρω από αυτό. Για τους δικαιούχους των κοινοτικών ταμείων τώρα και αυτών που την χάνουν κοινή διαχείριση, ιδιαίτερα για τη γεωργία και τους διαφθορτικούς τομείς, θεωρώ ότι θα πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν αυτό το σύστημα της έγκαιρης προειδοποίησης που να βασίζεται για αντίστοιχα και ισότιμα αναλυτικά κριτήρια σε όλες τις περιπτώσεις και ενώ σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει επίσης να δούμε με ποιο τρόπο συνδέονται οι απάτες με τα γενικότερα φαινόμενα διαφοράς τα οποία υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες. Θυμίζω το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2009 και το 80 σχεδόν της 100 των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι η διαφορά είναι βασικό πρόβλημα στη χώρα τους. Το 78% και το 76% πιστεύουν ότι υπάρχει διαφθορά και στα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα. Στα πλαίσια της καταπολέμησης τώρα της διαφθοράς και της καταπολέμησης της απάτης ε, προτείνω κάποια επιπλέον μέτρα. Τα μέτρα αυτά αφορούν αποτρεπτικές κυρώσεις κατάσχεση εν περιπτώσει ε, περιουσιών σε περιπτώσεις έκπληξης χρημάτων ή φορολογικών απατών όπως ακριβώς ε, προβλέπονται άλλωστε και στην οδηγία για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, την τρίτη στη σειρά. Θα πρέπει να γίνει επίσης και συγκεκριμένη αναφορά στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης που αφορά το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα είναι ένας επιπλέον μηχανισμός καταμέτρησης των επιπέδων διαφθοράς στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσιονομικού ελέγχου και συγκεκριμένα των προμηθειών, των κρατικών προμηθειών. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες της υπεύθυνε για την καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, Υπάρχουν μέσα στη διάθεσή μας τα οποία δεν χρησιμοποιούμε πλήρως για διάφορους λόγους και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στη Σύμβαση Αμοιβαίας Νομικής Συνδρομής όπως επίσης και στην Οδηγία Πλαίσιο για τις εντολές κατάσχεσης, προσωρινής κατάσχεσης και οικονομικών κυρώσεων. Θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης να προχωρήσει σε ε, μέτρα σχετικά ε, με τους αποκλεισμούς επαγγελματιών και επιχειρήσεων ε, από συμμετοχές σε περαιτέρω, σε επιχειρήσεις στο μέλλον. Η συμμετοχή κάποιων προσώπων τα οποία έχουν καταδικαστεί σε διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να αποκλείεται. Όλα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν και σε επιπλέον λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των παράνομων φορολογικών δραστηριοτήτων, μία πρόταση θα είναι το να αποκλείονται κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ε, καταδικαστεί στις χώρες τους, ακόμα και οι λεγόμενες εταιρείες offshore. Ζητάμε από το Συμβούλιο επίσης να κλείσει τη Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας με το Λίχτενστάιν γιατί έχει μπλοκαριστεί από ό,τι νομίζω και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης να ζητήσει από το Συμβούλιο να αποκτήσει εντολή για διαπραγμάτευση τέτοιων συμφωνιών με την Ανδόρα, το Μονακό και άλλες μικρές τέτοιες χώρες. στα πλαίσια πάντα των προσπαθειών καταπολέμησης των απατών και παρατυπιών, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η φορολογία. Τέλος, θα κάνω κάποιες γρατές προτάσεις σχετικά με τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση του θέματος προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οργανωμένο έγκλημα έχουν εμπλοκαριστεί από το Συμβούλιο οι προσπάθειες αυτές ήδη από το 2005. Α, είμαι σκιώδη εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη συγκεκριμένη έκθεση και γι' αυτό επέμεινα. Το καταλάβαμε, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Αντρέασεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ναι, και ο κύριος Σμιτ έλαβε το θάρρος ε, να μου απευθύνει δημόσια σε αυτή τη συνεδρία στη σχόλια. Ας απαντήσω κι εγώ. Εγώ ξέρω τι κάνω. Εσείς δεν ξέρετε τι κάνετε εκ μέρους των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Για να απαντήσω λοιπόν και στον κύριο, για να συνεχίσω μάλλον με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Μπονίτσι στον κύριο Ντί. Είπατε ότι μεταξύ αρνητικής και θετικής δήλωση ε, του αρνητικού και θετικού προσήμου το σημαντικό είναι ότι υπάρχει εξέλιξη. Σε αυτή την απάντηση όμω, εγώ θα σα πω το εξή: Ότι ο φορολογούμενο δεν είναι ικανοποιημένο με μια εξέλιξη και μόνο. Θέλει τα λεφτά που πληρώνει να δαπανώνται όπω πρέπει. Δεν τον ενδιαφέρει η εξέλιξη. Δεν είναι ζήτημα η εξέλιξη. Ζήτημα είναι να δαπανώνται τα χρήματα σωστά. Και αυτή είναι η δουλειά μου, κύριε Σμιτ. να προσέχω έτσι το τα λεφτά που δαπανάει η Επιτροπή να δαπανώνται σωστά. Για τον κύριο Κάλλας θα ήθελα να απαντήσετε στην ερώτηση που έθεσα νωρίτερα στον κύριο Σέμετα. Είχε μιλήσει η Επιτροπή πρώτη για μηδενική ανοχή στην διαφθορά. Τώρα μιλάτε για ανεκτό ποσοστό σφάλματος. Πώς έγινε και κατεβάσαμε τόσο τον πύχη. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Λυπάμαι που έφυγε ο εισηγητής. Αλλά υπάρχουν ισχυώδεις εισηγητές και υπάρχει φυσικά εδώ και ο Επίτροπος Κάλλας. Προσωπική μου άποψη είναι ότι οι απάτες δεν έχουν μειωθεί, αντίθετα έχουν αυξηθεί ουσιαστικά. Το πρόβλημα είναι η ικανότητα που θα πρέπει να έχουν τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά και θα πρέπει να είναι σε θέση η ΟΛΑΦ επίσης να τα ελέγχει αυτά τα συστήματα τα ελεγκτικά. Βλέπουμε ότι μέσω των απατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω του ελέγχου των δημοσιονομικών οδηγούμεθα στις βαρύτερες μορφές διαφθοράς που υπάρχουν στην Ευρώπη σήμερα και ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες. Οι δημόσιες προμήθειες και οι κρατικές προμήθειες είναι θα έλεγα παράδεισος και τρομερή ευκαιρία για τις μαφιόζικες οργανώσεις να κερδίσουν χρήματα. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Εγώ άκουσα την Τρίτη του Γενικού Γραμματέα, την απάντηση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είπε ότι υπάρχει μια διάκριση την οποία θα πρέπει να κάνουμε ανάμεσα στην παρατυπία και την απάνη. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην απάτη και τις παρατυπίες. Ξέρουμε επίσης τι σημαίνει διαφθορά. Και αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος μας να έχουμε περισσότερα στοιχεία γύρω από όλα αυτά. Ένα άλλο σημείο, ο κύριος Κάλλας δεν θα ασχοληθεί από εδώ και πέρα με το θέμα αυτό, αλλά μπορεί να μεταφέρει την ανησυχία μου σε αυτόν ο οποίος θα τον διαδεχθεί. Πέραν του ότι πρέπει να υποδεικνύουμε και να καταγγέλουμε δημόσια τα κράτη-μέλη τα οποία επανειλημμένα έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς και στις οποίες χώρες υπάρχουν σοβαρές απάτες ή έχουν σημειωθεί σοβαρές απάτες. Εσείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι στοχεύετε να κάνετε στα πλαίσια της αυτονομίας που έχετε απέναντι σε αυτά τα κράτη-μέλη. Ένα άλλο θέμα το συζητήσαμε ήδη στα πλαίσια της ακρόασης του Επιτρόπου Καγιάννη για το ε, Γαλιλαίο. Η οδηγία για τις κρατικές προμήθειες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και υπάρχουν και ε, σκοτεινές θα έλεγα περιοχές στα πλαίσια αυτής της οδηγίας που επιτρέπουν να μην αναπτύσσονται οι τάσεις για διαφάνεια με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε τους επόμενους μήνες να καταστήσουμε ικανή την ΟΛΑΦ να εργαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία, τουλάχιστον σε σχέση με το παρελθόν. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών οικονομικών βοηθειών και ε, κροών προς τις διάφορες χώρες είναι επαναλαμβάνω τρομερή ευκαιρία για ε, οικονομικά κέρδη από πλευράς του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος. Και το είπε και η κυρία Μακοβέ, η κυρία Γκρέσλε. Κύριε Πρόεδρε, τα ζητήματα που μας απασχόλησαν ε, θα ήθελα να τα συνεψίσω τόσο αν Νομίζω ότι μιλάμε τόσο ή άλλως για την ε, απαλλαγή του 2008. Ε, εν πάση περιπτώσει αυτός είναι αρμόδιος αυτή τη στιγμή, Επίτροπος. Δεν δε βγαίνω στα Ιταλικά. Ο κύριος Κάλλας ε, θα μας μιλήσει για την έκθεση Κοτσολίνο. Και μετά τώρα για το 2008 θα δούμε αν θέλει κάτι να προσθέσει. Τώρα μιλάμε μόνο για την έκθεση Κοτσολίνο, τίποτα άλλο. Κύριε Κάλλας, θα δώσετε απαντήσεις σε αυτά τα οποία τέθησαν. Πολύ σύντομα, δύο σημεία που επεσήμαναν τα μέλη της Επιτροπής σας. Και βεβαίως η διαφθορά σε οποιαδήποτε μορφή και να εμφανίζεται, ακόμη και υποψία, υποψία διαφθοράς, θα πρέπει να διαρευνάται. Αναμφίβολα δεν έχουμε αλλάξει στάση σε αυτό το θέμα και οποιαδήποτε παρατυπία ε, ε διαρευνάται. Μιλάμε για αποδεκτό προ το Υπό τον έλεγχο τη δική σα επιτροπή, πάντα σε εσά ερχόμαστε, υποβάλλουμε τα στοιχεία και εσεί τα κρίνετε και για το 2010 θα έχουμε τις πρώτες εκτιμήσεις αξιολογήσεις για την έρευνα, τις μεταφορές και τη γεωργία. Και την περιφερειακή ανάπτυξη, όχι τη γεωργία. Ε, συγγνώμη, όχι περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά υπαίθρου. Ε, και στο τέλος του χρόνου ο Επίτροπος θα έρθει με τα διοικητικά έξοδα και την απόδοση των λογαριασμών με διαφορετικά ποσοστά φυσικά και στους κινδύνους. Αυτή είναι η μεθοδολογία, μια μεθοδολογία και τίποτε περισσότερο. Οι παρατυπίες δεν είναι διαφθορά. Ε, είναι συνήθως καθυστερήσεις ως προς την υποβολή των αγράφων, ε, εκθέσεων κτλ. Που βεβαίως μπορεί πίσω από αυτές να υποκρύπτεται κάποια προσπάθεια διαφθοράς. Ε, γι' αυτό και τα ελέγχουμε πάντοτε. Να μην υπάρχει παραμικρή αμβολία σε αυτό. σε, κάποια, σε κάποιες παρατηρήσεις που είπαν ότι κέριο στοιχείο σε αυτήν την ιστορία, στοιχείο κλειδί είναι η συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ναι, όντως και εδώ έχουμε σημαντική βελτίωση γιατί πολλές φορές στο παρελθόν είχαμε ω προ την ανταπόκριση των κρατών μελών. Στέλναμε του φακέλου προ διερεύνηση στα κράτη-μέλη και πολλέ φορέ ούτε καν απαντούσαν στα αιτήματά μα. Ούτε μα λέγανε καν τι συνέχεια είχαν δώσει αυτά ε, τα αιτήματα. Τώρα με την νέα συνθήκη ορίζονται νέε υποχρεώσει για τα κράτη-μέλη και αντίστοιχε βέβαια δυνατότητε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για παρακολούθηση αυτών των υποθέσεων. Για το μισό-μισό, 50-50 που αναφέρθηκε, είναι βεβαίως καινοτόμο στοιχείο. Δεν ε, κέρδισε μεγάλη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη, αλλά πάντως μας ενθάρρυνε στις δραστηριότητες μας για ανάκτηση των κονδυλίων και στις προσπάθειές μας πάνω απ' όλα να εξασφαλίσουμε πως τα χρήματα δαπανώνται εκεί που πρέπει να δαπανηθούν. Φυσικά μπορεί να φτάσει η Επιτροπή μέχρι τη ε, διακοπή τη λειτουργία ενό προγράμματο ή και τη 100% ανακτήσεω θεωρητικά. Πάντω λειτουργεί το σύστημα όπω έχει με τι πιέσει αυτέ και θα πρέπει να διατηρηθεί και να δούμε τι αποτελέσματα φέρνει και περαιτέρω αν χρειαστεί κάποια άλλη ε, εξέλιξη. Για την διαφάνεια που έθιξε η κυρία Μακόβεϊ, πρέπει να σας πω ότι ε, με πιάνει μια νοσταλγία για τις ακροάσεις του 2004 που τις ε, ε, σχετικές ερωτήσεις για τη διαφάνεια τι απευθύνατε στον υποψήφιο, στην υποψήφια για την θέση αυτή και πρέπει να πω ότι από τις τότε απαντήσεις μόνο δύο χώρες είχαν δώσει λεπτομερείς καταστάσεις των ε, δικαιούχων. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα λοιπόν και είναι για όλες τις χώρες ε, οι καταστάσεις αυτές έτοιμες. Άρα μεγάλη αλλαγή βλέπω και ουσιαστική αλλαγή βλέπω προς τη συμπεριφορά των κρατών μελών με δημοσίευση από το 2009 δημόσια δημόσια κοινοποιούνται ε, δημοσιεύονται καλύτερα τα στοιχεία για όλα τα κράτη-μέλη. Ήταν βέβαια και ζήτημα μηχανογράφηση λίγο, γιατί υπάρχουν κάποια συστήματα δικά μας μηχανογραφικά, μέσα από τα οποία μπορείτε να περάσετε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε τα στοιχεία. Φυσικά αυτές οι εφαρμογές, οι ηλεκτρονικές, ε, μπορούν ε, να ε, βελτιωθούν ενδεχομένως για να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες. Αλλά το γεγονός είναι και μένει ότι δημοσιεύονται τα στοιχεία των δικαιούχων, τα, οι καταστάσεις των δικαιούχων και είναι προσβάσιμες στους πάντες. Για την κυρία Μακόβε επίσης οι διάφορες συμβάσεις που την ανησυχούν και που παρακολύουν τα κράτη-μέλη. Ναι, βεβαίω η νέα συνθήκη όμω μας δίνει νέες ε, δυνατότητες και η Όλαφ είναι παρούσα σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσει. πρωτοστατή θα έλεγα και με το Λίχτενστάιν και με τις ε, καπνοβιομηχανίε, που ξέρετε ότι είχαν μεγάλη σημασία και έγιναν πολλές ε, τέτοιε επαφές και δραστηριότητε και ως προς την αντιμετώπιση των τελωνιακών παρατυπιών δάσμο διαφυγής, ε, προβλήματα δηλαδή προς την καταβολή των δασμών που ε, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη, δυσκολία ως προς την πρόσβαση που μπορεί να έχουν τα κράτη-μέλη σε προβλήματα απάτης περί τους δασμούς όπου βεβαίως δραστηριοποιείται και το μεγαλύτερο ε, σε μεγαλύτερο βαθμό το οργανωμένο έγκλημα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσεκτική διερεύνηση είναι λεπτή δουλειά, περίπλοκη δουλειά. Η Όλαφ όμω μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει βοηθήσει πολύ τα κράτη-μέλη προσφέροντά του πολύτιμε πληροφορίε εκεί που είχαν ανάγκη για ε, συνεργασία. Και εγώ ίδιο επεσκέφθην ε, την, ε, τα γραφεία του στη Γερμανία. Ένας αγώνας ατέρμονος είναι αυτό, ένα αγώνα που πάντα μας φέρει αντιμέτωπους με μια νέα εξέλιξη, πάντα κάτι καινούριο προκύπτει, δεν σταματάμε ποτέ. Και φυσικά έχουμε τεράστια ευαισθησία ως προς την αξιοποίηση των κονδυλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα τα θεσμικά όργανα, σας διαβεβαιώ, ε, εξετάσουν με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα κάθε υπόνοια ακόμη παρατυπίας ή διαφθοράς. Ευχαριστώ πολύ. Α πάμε στην απαλλαγή 2008 τώρα. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο Κάλλα, θα παρακαλέσω τον κύριο Μπονίση εκ μέρου του ελεγκτικού συνεδρίου να μα πει αν έχει να προσθέσει τίποτε περισσότερο σχέση με αυτά που αρχικά. Είσαστε εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάλλας, έχετε το λόγο. Thank you very much. This is... Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για εμένα προφανώς δεν ξέρουμε, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Φαίνεται πως είναι η τελευταία φορά που είμαι ενώπιόν σας υπεύθυνος για την απαλλαγή και δεν θέλω τώρα να απαριθμίσω το σημαντικό έργο που έχουμε κάνει μαζί. Απλά να... Ξεχ... να θυμηθούμε το έργο που έχει γίνει από το 2005-2009 για τη μεταρρύθμιση της και την καταπολέμηση της απάτης. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα την αιτήσια έκθεση του 2008 να υπενθυμίσω τη γενική αντίδραση της Κομισιόν όπως εκδηλώθηκε το Νοέμβρη. Θεωρούσαμε πως η δήλωση εξοπιστίας του 2008 ήταν η καλύτερη που είχε γίνει ποτέ, αλλά βεβαίως σαφώς το ελεγκτικό συνέδριο μας λέει τι πρέπει να γίνει. Το μασικό μου μήνυμα άρα σήμερα είναι πως ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο ψηλό επίπεδο φιλοδοξίας. Να δώσω λοιπόν κάποια παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα να σας διαβεβαιώσω πως η Κομισιόν θα διατηρήσει το στρατηγικό στόχο να προσπαθεί για μια θετική διαβεβαίωση αξιοπιστίας καθώς πρόκειται για συλλογική απόφαση. Τίποτα λιγότερο δεν μπορούμε να αναμένουμε. Όπως άκουσα και ο κύριος Σεμέτα το ίδιο σας είπε για τα διαρθρωτικά ταμεία το βασικό πρόβλημα το οποίο παραμένει ε, φαίνεται πως αποδίδουν οι προσπάθειες της ε, Κομισιόν για την έκθεση αντικτύπου για τα διαστατικά ταμεία που θα υποβληθεί τον Φεβρουάριο ακριβώς για να μπορέσετε έγκαιρα να την εξετάσετε για να δείτε το χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος στα στηματα 2007 2007-2008. Εν πάση περιπτώσει, ο υποψήφιο Επίτροπος Χάν έχει καταστήσει και αυτός βασικό του μέλημα την καλύτερη διαχείριση. Είπε πως το ποσοστό στο 11% είναι καμπανάκι. Επίσης, τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με την Επιτροπή σας προσπαθούμε να τα τοπίσουμε την ευθύνη στα κράτη-μέλη, να αναλάβουν τις ευθύνε τους μάλλον. Παραδείγματο χάρη ο υποψήφιος επίτροπος ο κ. Λεβαντόφσκι ε, ε, αυτό το οποίο αναφέρονταν στην εκτεσύνδεση του 2008, ότι θα προτείνουμε δηλαδή ενίσχυση νομικού πλαισίου στον επόμενο δημοσιονομικό κανονισμό για ετήσιε ανακεφαλαιωτικές εκθέσει. Και νομίζω πω και το Συμβούλιο προ την ίδια κατεύθυνση κινείται. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να θεωρήσουμε αυτές τις συνοπτικές εκθέσεις αξιόπιστες. Επίσης θα πρέπει να δούμε οι πρωτοπόρες χώρες όπως η Ολλανδία και η Σουηδία να δώσουν κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για να ενισχυθεί η προσθέμενη αξία. Να σας πω επίσης πόσο ικανοποιημένος ήμουν που έλαβα από τους δύο υπουργούς αυτών των χωρών, τους υπουργούς οικονομικών επιστολές που δήλωναν πως ε, η πρώτη Επιτροπή Μπαρόζο οπωσδήποτε έχει βελτιώσει την διάθεση των κοινωτικών κονδυλίων και θα δούμε τι θα γίνει με την ψηφοφορία στο Συμβούλιο. Έλαβα λοιπόν αυτή την επιστολή όπου αναγνώριζαν το έργο μας και σαφώς έλεγαν πως ε, τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο βεβαίως. για να γίνουν ένα επιχειρησιακό έγγραφο οι εθνικές δηλώσεις. Επίσης, να σας πω πως σκοπεύουμε να βελτιώσουμε τις εσωτερικές λειτουργίες ελέγχου και θα ακολουθήσουμε όλες τις σχετικές στάσεις. Ο κύριος Σεμέτα θα είναι τώρα αυτός ο υπεύθυνο και θα αναπτύξει τον κεντρικό του ρόλο στο πλαίσιο το γενικότερο της ε, ορθής διοίκησης εντός της Κομισιόν για την διαφάνεια. Ο κύριος Μπαρόζο σε επιστολή του αυτό το μήνα στον κύριο Μπούζεκ, στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, είπε πως θα ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας και εγώ απευθυνα μία επιστολή προς τις τρεις επιβεβαιώντας πως η Κομισιόν είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο για να έχουμε ένα κοινό αρχείο λόμπι για να συμπεριλάβουμε και μια δήλωση από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για τα χρήματα που λαμβάνουν από τον κοινωτικό προϋπολογισμό. Το 2008 ήταν, είχαμε μια καλή δήλωση ε, αξιοπιστία, η καλύτερη που είχε γίνει ποτέ, αλλά βεβαίω υπάρχουν ακόμη τομεί που πρέπει να βελτιωθούν. Νομίζω πως και η, και Επιτροπή σας βεβαίω αξίζει εύσημα και ελπίζω πως θα συμφωνήσετε πως ε, πρέπει να δοθεί απαλλαγή στην Κομισιόν για το 2008 και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Πριν ε, δώσω τον λόγο στον κύριο Ριμπεράτσκι να υπενθυμίσω την έκθεση Κοντσολίνο πως ε, πρέπει να καταδεθούν τροπολογίες μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Παρακαλώ κύριε Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κάλλας, να κάνω ένα μικρό σχόλιο, καθώς πρόκειται για την τελευταία μας ακρόαση. Πέρασαν πέντε καλά χρόνια με τον κύριο Κάλλας ε, και εκτιμούμε το ότι πολλά έγιναν. Σημειώθηκε ορατή πρόοδος όμως έχω την εντύπωση πως ε, μας έδειξε ένα ωραίο διαγραμμά εδώ πέρα ο κ. Μπονίτσι που μιλάει για βελτιώσεις το 2005-2008, τέσσερα χρόνια και ότι είχαμε βελτίωση 9%. Σημαίνει αυτό πως η βελτίωση ετήσια είναι 2,5% το έτος. Οπότε έχουμε ακόμα πολλά να επιτύχουμε και θα μας πάρει 20 χρόνια με αυτό το ρυθμό. Και έχω την εντύπωση πως είναι λίγο μεγάλο αυτό το διάστημα. Ίσως θα έπρεπε να επιταχύνουμε κάπως ε, την ε, διαδικασία. Αυτή η, γενική μου παρατήρηση και έχοντα κατά νου αυτό το οποίο είπα για το να δείξουμε την εκτίμησή μας επί τη ευκαιρία να κάνω κάποια ερωτήματα στον κύριο Επίτροπο. Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, τα σφάλματα στα διαρθρωτικά ταμεία. Μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα και άμεσα βήματα τα οποία θα λάβει η Κομισιόν και έχει λάβει ήδη το 2009 για να μειωθεί αυτό το 11% που παραμένει εδώ και αρκετό καιρό. Το 11% δηλαδή κονδυλίων των διερθωτικών ταμείων που δεν έχουν διατεθεί σύμφωνα με τους κανόνες. Τι μπορεί να γίνει κατά την άποψή σας, αυτή την η πρώτη μου ερώτηση. Θα απαντήσω αμέσως ή να περιμένω με όλες τις ερωτήσεις. Τα διαφορετικά ταμεία, θυμάστε όλες τις ακροάσεις που κάναμε τα τελευταία χρόνια, είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί να μας ανησυχεί. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε τον τελευταίο καιρό πολύ προσεκτικά είναι βέβαια περίπλοκο το θέμα των διαφορετικών ταμείων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των προγραμμάτων κοινή διαχείρισης, γιατί εκεί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις και στον τρόπο με τον οποίο καλούνται να εφαρμοστούν. δεν έχουμε ακόμα απορροφήσει πλήρως και αξιολογήσει πλήρως τα ε, προγράμματα πλαισίου των παρελθουσών περιόδων Εκεί το ποσοστό λάθους ήταν πολύ υψηλότερο, τώρα είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα, πιο δυναμικά θα έλεγα, είμαστε και εμείς πιο ευέλικτοι και νομίζω ότι θα καταλήξουμε για την περίοδο μετά το 2006 και για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές με κάποια μέσα στη διάθεσή μας τα οποία θα δουν ότι το ποσοστό αυτό αποδεκτού λάθος θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Κάθε χρόνο εμείς ενισχύουμε και την ανάκτηση των ποσών στην οποία προχωρούμε και στην επιβολή των κυρώσεων. Αυτή η τάση είναι συγκεκριμένη πλέον τα τελευταία δύο χρόνια. έχετε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, όπου έχουν σταματήσει πληρωμές σε διάφορες χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και εκτός από τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, έχουμε και πιο συγκεκριμένες μεθόδους, χρησιμοποιούμε πιο συγκεκριμένες μεθόδους και για τους τρόπους ανάκτησης των ποσών τα οποία δεν έχουν σωστά δοθεί. για τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής έχουν φτάσει οι ανακτήσεις ποσών ε, άνα των 2,5 δις. Επίσης 1,5 δις ε, το ποσό αφορά ε, τις κοινωνικές πολιτικές και 1,7 δις τα διαρθρωτικά ταμεία. Μιλάμε τώρα για πολύ ψηλά ποσά τα οποία έχουμε, στα οποία έχουμε προχωρήσει στην ανάκτησή τους. Παρόλα αυτά και παρόλες τις μεθοδολογικές δυσκολίες οι οποίες εξοκολουθούν να υπάρχουν, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Και αυτό που επαναλαμβάνω έχει σημασία είναι ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη είναι πιο ευαίσθητα σε σχέση με το θέμα αυτό πλέον. Τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν πάρει έχουν εξαναγκάσει αν θέλετε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά με διαφορετικό τρόπο. Ελπίζω να οδηγήσει αυτό σε μείωση του ποσοστού λαθών και στα διαρθρωτικά ταμεία. Σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι, γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Θα ήθελα να μιλήσω για τα εσωτερικά συστήματα και πλαίσια ελέγχου. Είπατε ότι θα πρέπει οι προσπάθειες αυτές που γίνονται να αντικατοπτρίζουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων αυτών. Πότε θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάλυση κόστους και ωφέλους των ελεγκτικών αυτών ολοκληρωμένων συστημάτων. Κάτι το οποίο δεν είναι μόνο αριθμητικά στοιχεία τα οποία περιμένουμε, αλλά είναι κάτι που άπτεται των αρχών μας, θα έλεγα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντά ο κύριος Κάλλας. Εκεί όπου έχει υπάρξει τέτοια προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Οπότε για το κόστος του ελέγχου θα σας δώσω στοιχεία στο τέλος του 2010. Έχουμε να κάνουμε πάντως με μια μεγάλη γκάμα θα έλεγα απαντήσεων στην ερώτησή σας σε κάποιες ε, περιπτώσεις εκεί όπου υπάρχουν ε, συστηματικά προβλήματα θα έλεγα παρατυπιών και απατών εκεί το κόστος του ελέγχου είναι και αυτό ιδιαίτερα υψηλό. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε τέτοιες περιοχές ή σε τέτοιους τομείς να το πω καλύτερα. Μερικές φορές σε ορισμένα προγράμματα το κόστος ελέγχου μπορεί να φτάσει και το 30% του συνολικού κόστους. Ξέρω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, λέει ο κ. Μπράσκη. Πάντα για τον κύριο Κάλλας. Μιλάτε πάντα με πολύ ενθουσιώδη τρόπο για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Σε επίπεδο οικονομικό, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει τι ενέργειες έχει αναλάβει έτσι ώστε να ελέγχει πάντα τα χρήματα τα οποία δίδονται στις ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ οι οποίες δρούν, αναλαμβάνουν δράση σε τομείς χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Βοήθεια έχουν ανοιχτούς οικονομικούς λογαριασμούς θα έλεγα και ελέγχονται συστηματικά. Είχε συζητηθεί πριν μερικά χρόνια το συγκεκριμένο θέμα και είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία μικιό. Οι περισσότερες δρούν στον τομέα του περιβάλλοντος. Και στις περιπτώσεις αυτές οι αρμόδιοι γενικοί διευθυντές, διευθυντές και διευθύνσεις γενικότερα είναι αυτές οι οποίες αξιολογούν τις ΜΚΟ για το αν είναι επιλέξιμες να διαχειριστούν κοινοτικέ επιδοτήσεις. Η προσπάθεια αυτή είναι μια συνεχής προσπάθεια. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε βέβαια την τα πληροφορικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να συλλέξουμε τις πληροφορίες αυτές και να παρουσιάσουμε ένα κατάλογο των οργανώσεων αυτών οι οποίες χρησιμοποιούν κοινωνικά, κοινοτικά κονδύλια σε λίγους μήνες θα υπάρχει ένας τέτοιος ε, δημοσιευμένος κατάλογος. Αν και υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με το πώς ορίζουμε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Εντάξει, θα σταματήσω εδώ για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να θέσουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Κάλλας για τις απαντήσεις σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Γκρέσλα. Ευχαριστώ ως ε, αρμόδιο επίτροπο για τον ε, Όλαφ λόγω της... Ε, θα ήθελα να επισημάνω τη μεγάλη ευαισθησία που απαιτείται εδώ πέρα και μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα για το διορισμό του μεταβατικού διευθυντή που έγινε κατά παράβαση των διοργανικών δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το διορθώσετε αυτό. Δεν είναι θέμα παιχνιδιών μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αφορά την νομιμοποίηση των δραστηριοτήτων του Όλαφ. Είναι πολύ επίγον ζήτημα και οι γενικοί γραμματές Day είπε χτε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εγώ έχω πολλούς λόγους ανησυχίας. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω την Κομισιόν, τον Αρμόδιο Επίτροπο, επιτέλους να το πάρει σοβαρά αυτό το θέμα. Δύο θέματα τώρα στα οποία θα ήθελα μία απάντηση οι αρμοδιότητες σας αφορούν το προσωπικό και νομίζω πως από την ε, τελευταία αύξηση των ε, μισθών ε, που θα πάει τελικά στο δικαστήριο πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση του συστήματος υπολογισμού. Θεωρείτε πως θα πρέπει να υπάρξει ένας νέος υπολογισμός της ετήσιας αναπροσαρμογής. Αν δούμε τον τρόπο αυτό δεν νομίζω πως είναι πλέον διάφανης δεύτερον ένα παλαιό πεδίο μάχης τα χρήματα για τα οικονομά. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια έσοδα από πλευράς κομισιών για ενοικιασμένα κτίρια και η ε, Κομισιόν θεωρεί πως επειδή τις ανήκουν τα κτίρια, τις ανήκουν και τα έσοδα και εμείς ζητούσαμε να πηγαίνουν αυτά τα χρήματα στον ε, προϋπολογισμό και υποτίθεται πως ε, θα πήγαιναν για την επέκταση του γυμναστηρίου. Τι γίνεται λοιπόν, γιατί τελικά εκεί δεν πήγανε. Um, uh, Αυτή η ερώτηση για το οικονομά, για τα καταστήματα είναι εγγεγραμμένοι μας στον προπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθηθούν οι δημοσιονομικές διαδικασίες, είναι σαφείς οι κανόνες που πρέπει να τηρηθούν. Πρόβλημα δεν βλέπω εγώ. Ίσως θεωρηθεί παράδοξο το ότι προβλέφθηκε αυτό το ποσό αρχικά έξω από τον προπολογισμό, αλλά τώρα δεν υπάρχει αυτή η ανομαλία πλέον. Είναι μέσα στον προπολογισμό με απόλυτη διαφάνεια, σαφήνεια των κανόνων, τυπικότητα και ω εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για τη μεθοδολογία. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε τρία βασικά ζητήματα. Η μέθοδος ε, υπολογισμού των ε, μισθών και όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα βεβαίω, αλλά να σας δώσω το ιστορικό υπόβαθρο. Πρόκειται για μια πολιτική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών, των συνδικάτων, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ε, είχε προβλεφθεί ότι θα εφαρμόζεται πάντα η μέθοδος και ότι, είναι, ότι δεν θα αμφισβητηθεί εάν κάποιος πει ε, κάνοντας τους υπολογισμούς ότι τα αποτελέσματα δεν τον βρίσκουν σύμφωνο δεν μπορεί να ανατραπεί. Είναι μια απόφαση που λήφθηκε πριν από πολλά χρόνια, ήταν δύσκολο να ληφθεί και δεν μπορεί να ανατραπεί. Εάν όμως θέλει κάποιος από τους εμπλεκόμενους φορείς να μεταβάλει το σύστημα των πληρωμών, θα πρέπει να ανατρέξει στη μέθοδο αυτή και να την αναθεωρήσει. Ε, η μέθοδος ΔΕ δημιουργήθηκε προκειμένου να, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που θα προκαλεί η ένταξη των νέων κρατών μελών ως προς την πληρωμή των ε, μισθών που ήταν ταχύτερη στην ε, τιμαριθμική της εξέλιξη σε σχέση με κάποιων κρατών που φοβήθηκαν ότι μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ τη τιμαριθμικές αναπροσαρμογές στους μισθούς επιτροπής. Γι' αυτό κάποια κράτη-μέλη συμφώνησαν και οδήγησαν σε αυτό το μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο είναι υπαρκτό, το οποίο είναι εσωτερικό το οποίο υφίσταται και είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου, όπως σε κάθε χώρα ισχύει και δεν μπορεί κάποιος ξαφνικά να πει «Α, για κοιτάξτε, τώρα αυτό το μοντέλο μας βγάζει σαν αποτέλεσμα ένα αποτέλεσμα που δεν μας αρέσει και πολύ, είναι λίγο παράξενο». Δεν θα το εφαρμόσουμε λοιπόν το μοντέλο. Όχι. Το μοντέλο εφαρμόζεται, αυτή είναι η συμφωνία και με τα συνδικαλιστικά σωματεία και με τα κράτη-μέλη κτλ. Όπω συμβαίνει σε κάθε χώρα, πιστεύω και στη δικιά μου τουλάχιστον έτσι συμβαίνει. Και στη Γαλλία, φαντάζομαι, η οποία διαπραγματεύεται τώρα την καταβολή των σχετικών ε, ε, προσαρμογών ε, κατά επίπεδο 5% στου υπαλλήλου τη. Έτσι λοιπόν, εάν οι υπάλληλοι οι μισθοί μάλλον των υπαλλήλων ή των εκπροσώπων του δημοσίου τομέα, αν θέλετε, κάθε χρόνο εξαρτώνται από την πολιτική βούληση κάποιων, ε, προφανώς θα γίνει θα επικρατήσει το χάο. Δεν πρόκειται να βρεθεί λύση. Εάν θεωρούμε ότι ο μηχανισμό αυτός είναι καλός, ας τον αναθεωρήσουμε από την αρχή. Ας γυρίσουμε πίσω, ας βρούμε νέε διαδικασίες. Μόνο αυτό υπάρχει σαν λύση. Τα κράτη-μέλη έχουν βέβαια ε, λόγω βαρύνοντα, την υπόθεση αυτή είναι αυτό που διαθέτουν τα κονδύλια και αν θεωρούν ότι ε, έχουν εύλογα επιχειρήματα ότι αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί γιατί του χρόνου θα δώσει άλλο αποτέλεσμα η μέθοδος δεν θα, δώσει ε, του χρόνου την αριθμική αναπροσαρμογή δεν θα υπάρξει αύξηση των μισθών είναι σαφές αυτό από τα τωρινά δεδομένα τι θα κάνουμε λοιπόν τότε θα πούμε ότι α, όχι, δεν μα αρέσει η μέθοδο γιατί δεν προσφέρει την αριθμική αναπροσαρμογή προ τα άνω και άρα θα πρέπει να τη δώσουμε ούτω ή άλλω την προσαρμογή. Την αύξηση. Έχω πολύ έντονε μνήμε από τι δύσκολε εμπειρίε που είχα στη δική μου την πατρίδα πριν έρθω να λάβω αυτά τα καθήκοντα από τέτοιου είδου προβλήματα. Γι' αυτό επιμένω και επαναλαμβάνω και φωνασκώ ότι δεν πρέπει να ανατραπεί η μέθοδο κατά αυτόν τον τρόπο. Εάν δεν μα αρέσει η μέθοδο, πάμε να την αναθεωρήσουμε. Αλλά όταν υφίσταται η μέθοδο, όταν υπάρχει η μέθοδο, πρέπει να εφαρμόζεται. Δεν μπορεί κανεί να βγαίνει και να λέει Δεν εφαρμόζω τη μέθοδο τώρα που δεν με συμφέρει, που δεν μου αρέσει. Για δε την Όλαφ. Τα ξέρω όλα αυτά που λέτε και πολύ καλά, μπράβο. Αλλά δεν ξέρω από εδώ και μπρο τι να κάνω. Το 2005 ο κύριο Μπρούνερ ήταν ε, γενικός διευθυντής ήδη ένα χρόνο στη θέση αυτή. Είχε λοιπόν κάθε εξουσία και προνομία να αναλάβει τις ευθύνες και τις αποφάσεις που χρειάζονταν. Εγώ χωρίς να είμαι δικηγόρος βλέπω, διαβάζω αυτά τα νομικά κείμενα και τα ψηλά γράμματα και όλες αυτές τις παρατηρήσεις τις τόσο περίπλοκες. Ερωτώ λοιπόν, εγώ τι να κάνω από εδώ και μπρος. Δυστυχώς απεδίωσε ο κύριος Μπρίνερ. Ε, πρέπει λοιπόν να βρεθεί κάποιος μηχανισμός να εξασφαλιστεί η διαχείριση, η διοίκηση του οργάνου άπαξ και απεβίωσε ο, ο, ο Γενικός Διευθυντής, πρέπει αυτός που ορίζεται δυνάμει και τον κανόνα του 2005 ήδη ω υπεύθυνο αναπληρωτή κλπ. να συνεχίσει τη δουλειά αυτή για να ξεκινήσει μια διαδικασία ε, για, το, ε, ε, για διαγωνισμό, για την προκήρυξη της θέσης γενικό Διευθυντή. Εάν έχει κάνει άλλη λύση, ταχύτερη για την αντικατάσταση του εκλειπώντο, πολύ ευχαρίστω. αλλά σα διαβεβαιώνω δεν θα είναι ταχύτερη, γιατί χρειάστηκε ένα χρόνο για να βρεθεί και να προχωρήσει η διαδικασία ε, για, το διορισμό του κυρίου Γκρίνερ. Θα ήταν εύκολο αν συμφωνούσαμε μεταξύ μα τα θεσμικά όργανα, αλλά δεν συμφωνούμε εύκολα μεταξύ μα και γι' αυτό και θα καθυστερήσει η διαδικασία τη προκήρυξη τη νέα θέση. Εδώ μεταξύ, τι γίνεται, Όλεφ. ποιο έχει την ευθύνη, ποιο την καθοδηγεί. Εγώ, ω μάνατζερ βλέποντά το, λέω δεν υπάρχει άλλη λύση μόνο αυτός ο οποίος ήδη με βάση την απόφαση της Επιτροπής του 2005 είναι αναπληρωτής και δυνάμει βέβαια και τις προτάσεις του τότε Γενικού Διευθυντού έχει οριστεί ως αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντού σε περίπτωση κολλήματος ή απουσίας. Εγώ πρακτικό πώ. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί η απουσιας εγω πρακτικός πως δεν χωρί κάποιον ολαφ χωρίς καποιον επικεφαλής που θα την καθοδηγεί, που θα την διευθύνει. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση τώρα. Ή πρέπει να βρούμε, να προκαλέσουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού, να διορίσουμε τον ε, αντικαταστάτη μέσα σε μια διοργανική διαδικασία που θα κρατήσει ένα χρόνο. Οπότε τι κάνουμε μέχρι τότε. Ή προχωρούμε. Όπως είπα, η διαδικασία κρατάει πολύ καιρό. Και πρέπει μέχρι τότε να βρούμε μία λύση. Αυτό λέω εγώ. Αλλά βέβαια ο κόσμος των νομικών είναι πολύ περίπλοκος και ίσως δεν μπορεί ένας απλοϊκός οικονομολόγος να καταλάβει όλα αυτά τα λεπτά ζητήματα και τις αποχρώσεις τις νομικές. Ευχαριστώ κυρία Αντρέασεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στις απαντήσεις τις οποίες δώσατε στις ερωτήσεις μας υπήρξε μια ερώτηση για τα υψηλά ποσοστά στην Ισπανία Υπάρχουν κάποιοι τομείς και εδώ έχω λάβει πολλά παράπονα από τους φορολογούμενους ότι υπάρχει τρομερή διαφθορά στον τομέα της πολεοδομίας στην Ισπανία. Γιατί να συνεχίζουμε να επιδοτούμε περιοχές στις οποίες υπάρχει τόσο υψηλό ποσοστό διαφθοράς, ποιος ο λόγος. Χθε η Γενική Γραμματέας, η κυρία Κάθιντεϊ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε ότι υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφορά των επιτρόπων. Εμείς πέρυσι είχαμε συζητήσει μια έκθεση με πολλές συστάσεις στο εσωτερικό της. Την έκθεσή μας θα αντιλάβετε υπόψη σας σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αναθεωρήσετε κατά συνεπία πέρα τον κώδικα συμπεριφοράς. Επίσης η κυρία Ντέι είπε ότι κάποιες αλλαγές σχετικά με τον κανονισμό τον υπαλληλικό θα αφορούν μόνο τις εξωτερικές υπηρεσίε. Αυτό ισχύει ή οι αλλαγέ θα αφορούν το σύνολο των υπαλλήλων. Για την Ισπανία εμείς διακόψαμε πέντε λειτουργικά προγράμματα και υπάρχουν ε, και κάποιες άλλες μορφές ελέγχου οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξη. Η Όλαφ εξετάζει όλα αυτά τα θέματα, είναι σοβαρά Και υπάρχει σοβαρή συνεργασία επίσης ανάμεσα στις ισπανικές αρχές και στις δικές μας αρχές, στις δικές μας υπηρεσίες. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε μόνο την περίπτωση της Ισπανίας. Δεν θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την Ισπανία. Υπάρχουν διακοπές προγραμμάτων και έχουμε ζητήσει 200 εκατομμύρια πίσω από την Ισπανία και έχουν σταματήσει επαναλαμβάνω πέντε προγράμματα. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες όμως. Γενικά οι Ισπανικές αρχές από ό,τι φαίνεται είναι σε θέση να διαχειριστούν το πρόβλημα. Η Ισπανία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα βέβαια και δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για όλες τις μικρότερες και μεγαλύτερες τοπικές κοινότητες για τον κώδικα συμπεριφοράς. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Πάντα μπορούμε να ρυθμίζουμε στις λεπτομέρειες τα κείμενα αυτά τα οποία διέπουν τη λειτουργία μας και την καθημερινή μας ζωή. Ένα τέτοιο κείμενο, ακριβώς επειδή είναι ιδιαίτερα σύνθετο, δεν θα είναι ποτέ τέλειο. Και ένα τέτοιο κείμενο θα τρέχει συνέχεια πίσω από τις εξελίξεις. Ήδη από το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός διοργανικού οργάνου εμπειρογνωμόνων που θα εξετάζει τα θέματα ε, της σύγκρουσης συμφερόντων, της σύπτωσης οικονομικών συμφερόντων κτλ. Όλα αυτά σε επίπεδο λεπτομεριών είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθοριστούν γραπτός. Η πρόταση που είχε γίνει τότε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απερίφθη από τα άλλα όργανα. Παρ' όλα αυτά δημιουργήσαμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια ομάδα δεοντολογίας η οποία εξετάζει τις περιπτώσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται, ιδιαίτερα για τους υψηλόβαθμους υπαλλήλους. Είναι ένα μεγάλο κείμενο αυτό και έχουμε ολοκληρώσει και μια μελέτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτός από τον κώδικα συμπεριφορά που ονομάζεται επαγγελματική δεοντολογία των, ε, αξιωμα... των δημοσίων αξιωματούχων σε ευρωπαϊκά όργανα. Αλλά δεν αφορά βέβαια, είναι γενικότερο το κείμενο, δεν αφορά μόνο τους ευρωϊπαλλήλους, αλλά και τους υπαλλήλου των δημοσίων υπηρεσιών και κάναμε συγκρίσεις και είδαμε ότι έχουμε περάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας. Και ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοιου είδους ρυθμίσεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Παρ' όλα αυτά η νέα Ευρωπαϊκή θα συζητήσει ένα νέο κώδικα συμπεριφοράς και θα λάβει υπόψη τις ε, ε, παρεμβάσεις όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων μεταξύ των οποίων και της Επιτροπής σας. Οι εξωτερικές δράσεις. Είναι δύο διαφορετικά θέματα εδώ. Υπάρχει μια άμεση ανάγκη να ρυθμίσουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και να την καταστήσουμε ικανή να λειτουργήσει με την καινούργια της μορφή και υπάρχει ένα πακέτο αποφάσεων οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν το ταχύτερο δυνατόν για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Δεν έχουμε όμως καμία πρόθεση εμείς να αναθεωρήσουμε σε βάθος τον υπαλληλικό κανονισμό. Κάποιες λεπτομέρειες και κάποια θέματα θα τεθούν σε συζήτηση και σε επίπεδο επίσης δημοσιονομικό, γιατί ένα βασικό θέμα παραμένει πάντα το δημοσιονομικό. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόγραμμα για μία σε βάθος αναθεώρηση του υπαλλολικού κανονισμού. Ο κ. Κατζημαρκάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω και εγώ με τον εισηγητή Πράγματι, έκανε μια στροφή ο κύριος Κάλλας, εισήγαγε μια αλλαγή. Τα νούμερα συνεχώς βελτιώνονται, είναι επίτευγμα, είναι ιστορικό. Νομίζω πρέπει να το πούμε μια που είναι η τελευταία μας συνεδρίαση μαζί του. Και βεβαίως αυτό εξαρτάται και από το τι έκανε το Κοινοβούλιο εδώ πέρα και το πώς θα συνεχίσουμε το Κοινοβούλιο έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην αλλαγή αυτή. Οπότε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Λιμπεράτσκι είναι αξιοσημείωτο. Πρέπει να το, να το εξετάσουμε γιατί αν δούμε τι, πώς συμπεριφερόμαστε ένα στον άλλον για το εάν θα υπάρξει απαλλαγή ή όχι τότε νομίζω μπορούμε να μιλήσουμε και για τα μεγάλα πράγματα. Δηλαδή ότι να χτυπάμε συνέχεια τα κράτη-μέλη και λέμε αυτά φταίνε, και άρα σας παίρνουμε κρατάμε σε ομοιρία την Κομισιόν δεν είναι έτσι με ενδιαφέρει η άποψη της Κομισιόν γιατί έχει εμπειρία αλλά πρέπει να επανεξετάσουμε θεμελιωδώς το ε, εάν ε, πρέπει να δώσουμε απαλλαγή σε μια Κομισιόν η οποία πλέον δεν είναι εν ενεργεία γιατί πάντα για το παρελθόν μιλάμε. Και πέρσι δώσαμε απαλλαγή γιατί είχαμε μπροστά μα συνθήκη Λισαβόνας και πρέπει να είμαστε πολιτικά ορθοί. Τώρα που ξεκινάει από την αρχή κομισιόν πρέπει να πούμε τα πράγματα καθαρά. Δηλαδή να δούμε το τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως κομισιόν οι ίδιοι και είχαμε αυτή την εβδομάδα μια πάρα πολύ άσχημη ή τέλος πάντων μια σαφή έκθεση από τον κύριο ε, τον κύριο Εγκβέρτα για τις εξωτερικές ε, δραστηριότητες. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Κομισιόν, τι μπορεί να κάνει για τον Όλαφ. Ε, είπατε μόνο σας πως ξέρω τι πρέπει να κάνω, πρέπει να το κάνουμε. Να δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τις δραστηριότητες του κυρίου Κρατά δεν ξέρω πώς έκανε περισσότερα από αυτά τα οποία το επιτρέπονταν. Θα αναφέρω τώρα δύο παραδείγματα στα οποία είστε υπεύθυνοι ως Κομισιόν και εμείς εξετάζουμε ως Κοινοβούλιο τι κάνετε. Η ΜΚΙΟ. Μας γράψατε εδώ πέρα ένα γράμμα προς τον πρόεδρό μας, ευγενικό, αλλά κατά βάση μας λέτε εδώ πέρα, κάντε το μόνοι σας. Πατήστε εκεί με το ποντίκι, είναι οι βάσεις δεδομένων ελεύθερες Έχουμε ζητήσει πολλές φορές ως Κοινοβούλιο να δείτε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι σωστό να περιμένουμε να έρθει νέος επίτροπος που αναγκάζεται επειδή θεωρεί ότι έχει μπροστά του τις Κροάσεις να δώσει απάντηση. Και αυτή η δουλειά έπρεπε να έχει γίνει από κάτι υπαλλήλους κομισιών. Πληρώνονται από ό,τι βλέπουμε στις εφημερίδες οπότε μπορούν να το κάνουν. Υποθέτω πως εδώ πέρα κρύβεται η πολιτική. Δεν θέλετε να μας πείτε ποια λεφτά δίνετε σε ποιους. Στο περιβάλλον ε, ζητήσαμε και εκεί πέρα πληροφορίες και λάβαμε πληροφορίες. Δηλαδή ότι υπάρχουν ΜΚΟ που είναι ενεργές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 60% του προπολογισμού είναι επιδότηση. Δείτε το. Στην, ε, στην counterbalance στην ιστοσελίδα τους. Ε, δεν είναι δυνατόν να τους πληρώνουμε και από πάνω. Και να μην ξέρουμε τι είναι. Δεύτερο παράδειγμα, οι εκτελεστικές ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Είχαμε εδώ πέρα μια πολύ καλή ανάλυση. Ήμουν συνυπεύθυνο και εγώ για μια τέτοια υπηρεσία. Γνωρίζω πως είναι καλό καλή αναλογία κόσοφέλους ε, γιατί έχουμε συμβασιούχου και κοστίζουν λιγότερο. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό το οποίο δεν γίνεται είναι το εάν οι στόχοι που ορίζουμε εμείς ως πολιτικοί εκπληρώνονται. Κοιτάτε εάν κάνουν τη δουλειά τους μόνο, δηλαδή εάν έχουν δαπανηθεί σωστά τα χρήματα. Για τους πολιτικούς στόχους δεν το αναλύεται. Αυτό ισχύει σε πολλές ε, περιπτώσεις. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια. Δεν έχει νόημα λοιπόν να ε, είμαστε ευγενικοί. Λόγω των ιστορικών επιτευγμάτων του κύριου Κάλλας έχω μια τέτοια τάση, αλλά η νέα Κομισιόν πρέπει πραγματικά εδώ πέρα, στην οποία θα ανήκετε κι εσείς, να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και το λέω ξεκάθαρα. Παρατηρήσαμε στις ακροάσεις πως γίνεται όλο και πιο προεδρικό το σύστημα. Όλα παραπέμπονται στον πρόεδρο. Εντάξει. Αλλά και ο ίδιος, άρα πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Να λάβει περισσότερες ευθύνες. Και ε, θα το συζητήσουμε αυτό ανοιχτά και χαίρομαι που έχουμε εδώ πέρα τον νυν αντιπρόεδρο και στο νέο σώμα των επιτρόπων θα μπορέσει να τα μεταφέρει αυτά γιατί Είχαμε κάνει μια ανάλογη ανατροπή στο Κοινοβούλιο πριν από λίγα χρόνια και πρέπει να κινηθούμε ξανά προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ για τις μη κυβερνητικέ οργανώσει. Μπορώ να σας συστήσω να τις προσκαλέσετε εδώ, να ακούσετε τι γνώμη έχουν να σα πούνε ποιο είναι υπέρ και ποιο είναι κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να του προτείνετε να σταματήσει η χρηματοδότηση για τις περιβαλλοντικές ε, ενώσεις, παραδείγματι, που είναι οι πιο αυστηρές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε εκεί πώς θα αντιδράσετε και πώς θα αντιδράσουν. Βεβαίως, ξέρουμε ότι είναι αυτό, ότι έτσι συμβαίνει. Εγώ όμως λέω το εξή: Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. Ποιος τι ποιος χρηματοδοτεί. Χρειαζόμαστε την άποψή τους. Χρειαζόμαστε τη δική τους τοποθέτηση. Ναι, άρα πρέπει να τις χρηματοδοτούμε. Βεβαίως, στον χώρο του περιβάλλοντος μπορεί κάποιες από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να μην εκδηλώνουν <clears throat> το ενδιαφέρον τους για το ίδιο σαφείς στόχους όσο εμείς. πάση περιπτώσει που να μην συμφωνούμε. Είναι όμως λεπτό το ζήτημα. Εδώ στην Επιτροπή μας πρέπει από μερικά χρόνια στην Επιτροπή σας που το συζητήσαμε και σας είχα δώσει και τις σχετικές απαντήσεις. Όπως και εγώ και τα σχετικές υπηρεσίες ε, τις δίνουν. Ε, εμείς δεν χρηματοδοτούμε μια μη κυβερνητική οργάνωση μόνο και μόνο για να υπάρχει. Χρηματοδοτούμε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Σχέδιο το οποίο ακολουθεί κανόνες, στόχους, δημοσιονομικό έλεγχο, λογιστικό έλεγχο, μερικές φορές αποδείχθη ότι δεν ήταν και τόσο ε, επιτυχής πάντα η επιλογή. Δηλαδή μερικές φορές τα χρήματα, τα χρήματα πήγαιναν σε μια μη κυβερνητική οργάνωση μόνο και μόνο επειδή υπήρχε και όχι σε κάποιο σχέδιο. Έστω. Αλλά είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό και σοβαρό. Ποιο θα ορίσει ποια είναι η μη κυβερνητική οργάνωση. Λέτε ότι διαρκώ τάσσονται κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά είναι οι περισσότερε είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώ επικριτικά στέκονται απέναντι στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνε, διατάξει κτλ. Άρα πρέπει να μιλήσουμε διαφορετικό ε, πνεύμα για την διαφάνεια και την καταπλέμιση διαφορά κτλ. Το Μητρό, ναι βεβαίω είναι κάτι το καινούριο, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή χρειάζεται χρόνο να ρονταριστεί και ξέρω ότι ένα από του ε, διαδόχου μου θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό των μη κυβερνητικών οργανώσεων και την εγγραφή του στο καταστατικό, στο μητρό αυτό. Θα χρειαστεί όμω χρόνο. Τώρα, για του εκτελεστικού οργανισμού, Υπάρχουν δύο τύποι εκτελεστικών οργανισμών που είναι αφενό μεν οι ρυθμιστικοί, υπό το δικό σα έλεγχο, οι περισσότεροι, 23 των αριθμών, δεν απατώμε, και οι εκτελεστικοί είναι που είναι ε, που υπάγονται στι ε, υπηρεσίε επιτροπή όπου έχουμε εμεί την ευθύνη. Και εκεί δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το ποιο έχει ποια ευθύνη. Και υπάγονται και στο δημοσιονομικό έλεγχο και στην αξιολόγηση των πολιτικών, ε, του προϊόντος τους πολιτικός. Υπήρξε περίπτωση ε, ε, τέτοιου οργανισμού που έκλεισε όταν εξέπνευσε ο λόγος ύπαρξής του. Εγώ προσωπικώς υπό την ευθύνη μου είχα μία, έναν εκτελεστικό και τρεις ρυθμιστικούς οργανισμούς. Είχα μάλιστα και την πρωτοβουλία να παραπέμψω το θέμα στο ελεγκτικό συνέδριο. Ξέρω ότι δεν άρεσε σε ορισμένους αυτή η πρωτοβουλία. Ε, αλλά σας διαβεβαιώ ότι αυτή είναι η θέση μου πάντα, να είμαι δηλαδή ιδιαίτερα προσεκτικός στην ε, άψογη διαχείριση. Επίσης, από τα όσα συστήθηκαν και από την τελευταία θητεία, Βλέπω ότι τα προβλήματα πιο πολύ εμφανίζονται σε επίπεδο ρυθμιστικών οργανισμών, όπου επικρατεί διαφορετική απαλλαγή, υπάρχει σύστημα χωριστή απαλλαγή. Αλλά αν κανεί πει, κοιτάξτε κάτι δεν πάει καλά, γιατί δεν πάει καλά, υπεύθυνο πάλι είναι ο Επίτροπο. Στην τελευταία ανάλυση εσείς συστάτε και την απαλλαγή της Επιτροπής και χωριστά τους 20 ε, τόσους οργανισμούς. Ξέρω ότι επιμελητιακά ίσω είναι δύσκολο να οργανωθεί αυτό και δεν μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα την ακρόαση όλων των οργανισμών και τη Επιτροπή, αλλά πάντω ε, περισσότερου του ενό μπορείτε να δείτε ταυτόχρονα. ξέρω ότι ε, γενικά και στην Επιτροπή άλλος έχει ο καθένας έχει το δικό του στυλ και άλλος έχει πιο πολύ την πρωτοβουλία, άλλος λιγότερο, αλλά εγώ προσωπικώς για τον προϋπολογισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού ήμουνα άτεκτος και σε αυτό είχα και την υποστήριξη του Προέδρου. Χωρίς να μπορώ να ισχυριστώ ότι υπήρξε παρενόχληση από κάποιον άλλον ε, συνάδελφο. αντιθέτω, από κοινού συνεργαστικά με σε πνεύμα αγαστό και αν έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αγιάλα, Σέντζαρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από οτιδήποτε άλλο θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση μετά από την παρέμβαση τη κυρία Αντρέασεν για την Ισπανία. Ίσως δεν είναι απόλυτα ενημερωμένη η κυρία Αντρέασεν γιατί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ισπανία βρίσκεται και η Μεγάλη Βρετανία. Εγώ προσπαθώ να βρω κάποιες λύσεις όπου αυτό είναι δυνατό στη χώρα μου και θα πρέπει επίσης να ζητήσουμε και από τις Βρετανικές τράπεζες να μας πούν αν είναι αυτές που προκάλεσαν ένα μεγάλο ποσοστό της κρίσης το οποίο συναντάμε στην Ισπανία. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον κύριο Κάλλας για την νέα του εντολή τη στιγμή που ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τον διάλογο, τον καρποφόρο τον οποίο είχαμε μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να ζητήσουμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικές με την, θα έλεγα, με την κληρονομιά την οποία έχουμε πλέον μπροστά μας ε, σχετικά με τις ελεγκτικές διαδικασίες. Μας είπε ο κύριος Μπονίτσι το τι γίνεται με τις διαδικασίες ελέγχου σε τομείς όπως η Γεωργία. Εκεί ο έλεγχος είναι σχετικά αποτελεσματικός. Επίσης μας μιλήσατε για τους ελέγχους στον τομέα της συνοχής. Εκεί είπαμε ότι το κόστος των ελέγχων είναι και χαμηλότερο από ό,τι συνήθως σε άλλους τομείς. Απ' την άλλη είπατε ότι σε ορισμένα προγράμματα το κόστος του ελέγχου ανέρχεται περίπου στο 30%. Ως εκ τούτου τι ακριβώς πρέπει να καταλάβουμε από αυτά τα τρία στοιχεία. Από ό,τι βλέπω η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς σαν Ευρωβουλευτές ασκούμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι τμήμα της δημοκρατίας και της ελευθερίας έκφρασης. Το μόνο που μπορούμε να απαιτήσουμε και να ζητήσουμε είναι να υπογραμμιστεί η ευρωπαϊκή πρωτιστέμενη αξία. Θα πρέπει σίγουρα να ε, συνεργαστούμε με καλύτερο τρόπο με τις μη, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι κριτικές τις οποίες ασκούν αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι πολλές φορές ε, ε, επικοδομητικοί. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε σε σχέση με τις ΜΚΟ. Προφανώς υπάρχει ένα θέμα διαφάνειας, αλλά επειδή υπάρχει ένα θέμα διαφάνειας δεν σημαίνει ότι πρέπει να διακόψουμε τη συνεργασία μαζί τους. Το θέμα της ΟΛΑΦ είναι κάτι το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα κύριε Κάλλας. Όπως και εσάς άλλωστε όπως είπατε. Εγώ νιώθω συνυπεύθυνη σαν βουλευτής στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί δεν μπορέσαμε να προβλέψουμε ένα σύστημα το οποίο να επιτρέψει ε, την συνέχιση της διαδικασίας λειτουργίας της ΟΛΑΦ μετά τον ατυχή και απρόβλεπτο ε, θάνατο του προηγούμενου διευθυντή. Υπάρχει μια έλλειψη εδώ ε, θεσμική και ο νέος υπεύθυνος παίρνει κάποιες αποφάσεις χωρίς να έχει ελέγξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πραγματική πολιτική ανεξαρτησία του συγκεκριμένου προσώπου. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Ντεμάγκιστρης, είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει και επί τη βάση της γνωμοθέτησης της ε, νομικής επιτροπής ε, το τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να οργανωθεί μια ακρόαση με το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή, αντικαθιστώντας ε, τον κύριο Μπρούνερ. Κύριος Κάλλας. Θα πρέπει να είσαστε σύντομοι γιατί έχουμε άλλο ένα θέμα και πρέπει να τελειώσουμε στις 12. Ευχαριστώ. Για να απαντήσω ως προς την ανεξαρτησία της Όλαφ. Και μια και ούτως άλλως ασχέθηκε νωρίτερα όλη αυτή η υπόθεση. Η ανεξαρτησία λειτουργικά, σε λειτουργικούς όρους της Όλαφ, ποτέ αυτά τα πέντε χρόνια δεν τέθη ένα αμφιβόλο. Πριν από κανένα δύο χρόνια είχαμε μια συζήτηση που κατέληξε λόγω κάποιου προβλήματο που είχε εμφανιστεί το 2004, τώρα ότι ξεκινήσαμε. Ήταν τεράστιο θέμα, καυτό θέμα στην επικαιρότητα. Και ε, ψάχναμε τον τρόπο να βρούμε πώ θα λειτουργούσε η Όλαφ χωρί κανείς να μπορεί να παρέμβει στις ερευνέ τη. Έγινε η ακρόαση και εξετάστηκε ει βάθο όλο αυτό το θέμα, όλα αυτά τα θέματα και καταλήξαμε τελικά ότι δεν παραβιάστηκαν ποτέ οι κανόνες. Και βεβαίως και τα ε, ποπτικά συμβούλια είναι πολύ ε, σοβαρά στην έρευνά τους. Αν ποτέ υπάρξει η παραμικρή αμφισβήτηση βεβαίως θα την εξετάσουν. Εγώ σημειώνω μόνο ότι πάντοτε τηρούσα απαρέκλητα τη γραμμή του απόλυτου σεβασμού Τη ανεξαρτησία τη Όλαφ και δεν πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει, ούτε θα ήθελα να αλλάξει. Άουντι για την τελευταία παρέμβαση. Κύριο Σοντζή, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να πω πόσο πολύ θα μας λείψετε, γιατί εκτιμώ ιδιαίτερα τις ε, ικανότητες σας, αλλά και ως βουλευτής εκτιμώ και την υπομονή σας και την αποφασιστικότητά σας και την ηρεμία σας. Και πολύ περισσότερο γιατί όταν σας βλέπουμε εδώ μέσα στην αίθουσά μας να διαβάζετε τις υπηρεσίες, τα έγγραφα που σας ε, δίνουν οι υπηρεσίες σας στην αρχή φαινόταν σαν να βαριέστε λίγο. Τώρα βλέπω όμως να έχετε φτάσει σε επίπεδα δεξιότητα. Είσαστε ένας βιρτουόζος και σας ευχαριστώ πολύ για όσες προσπάθειες καταβάλατε για την απαλλαγή και πάνω απ' όλα σας συγχαίρω που σας επέλεξε το κράτος μέλος σας ως ψήφιο επίτροπο. Και το ερώτημά μου είναι πολύ σύντομο κύριε επίτροπε, το ίδιο από αυτό που υπέβαλα και στον ε, καθηγητή Μπονέτσι, πώς δηλαδή διαβάζετε εσείς την έκθεση του λεκτικού συνεδρίου για το 2008. Είπαμε ότι για χρόνια είχαμε αρνητικές ε, δηλώσεις αξιοπιστίας. Εγώ ρώτησα τον κύριο Πονίτσα, είναι θετική η τωρινή, μου απάντησε ναι, έχουμε εξελίξει θετικέ και τα λοιπά, όλα πάνε καλύτερα, αλλά ως ελεκτής δημοσιονομικός, ήσασταν επικεφαλής ελεκτικών υπηρεσιών πρέπει να είναι ο δημοσιονομικό ελέγκτης σε θέση να πει δίνω θετική ή αρνητική ή θετική με επιφυλάξει δήλωση αξιοπιστία. Γι' αυτό λοιπόν και ως μέλος βεβαίως της Επιτροπής Συλλογικού ε, Οργάνου αλλά και ως θεματοφύλακος των συνθήκων και δυνάμει πάνω απ' όλα του άρθρου 248 που καλεί την Επιτροπή να τοποθετείται, όχι απλώς να δίνει κάποια γνωμοδότηση και γιατί όταν ήμουν εγώ εισηγητής έπρεπε να εξετάσουμε αν θα αναβληθεί η απαλλαγή του προπολογισμού. Τελικά είπαμε, προτείναμε στο Κοινοβούλιο να δεχθεί την απαλλαγή, αλλά μέσα σε δεδομένα πολιτική πολιτικών ε, αντιπαραθέσεων ε, δύσκολα γιατί θυμάστε είχαμε τις ευρωεκλογέ μπροστά μας. Τώρα όμως είμαστε σε διαφορετικές συνθήκες και πολιτικά διαφορετικές με στην αρχή μιας θητείας και ρωτώ εάν εσείς αυτή την έκθεση τη βλέπετε ως θετική ε, δήλωση αξιοπιστίας ή αρνητική. Κάποιος υπάλληλο μου έλεγε πρόσφατα ναι, το κοινοβούλιο δαγκώνει πολύ, αλλά δεν, ε, γαυγίζει πολύ αλλά δεν δαγκώνει. Σήμερα όμως μπορεί τελικά αυτές οι συζητήσεις να μας οδηγήσουν σε μια κατάσταση στην οποία πράγματι θα πρέπει να γνωρίζουμε εάν η δήλωση αξιοπιστίας είναι θετική ή μη. Εσείς λοιπόν πώς ε, ερμηνεύετε την πρόταση του ελεκτικού συνεδρίου για το άρθρο που αναφέρατε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά πολλά καλά λόγια πρέπει να πούμε και για τον καθηγητή τον κύριο Μπονίτσι που έπαιξε κέριο ρόλο για να γίνει αυτή η δήλωση εξοπιστίας πιο ευανάγνωστη και κατανοητή. Και υπ' αυτή την έννοια είχαμε ένα κοινό συμφέρον να βελτιωθεί δηλαδή η οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση και το ελεγκτικό συνέδριο μας βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε το κείμενο αυτό βεβαίως αντικατοπτρίζει την κατάσταση και οι δύο-τρεις σελίδες είναι όπως πρέπει. Το μόνο πρόβλημα είναι πως η συνθήκη απαιτεί το ελεγκτικό συνέδριο να δώσει διαβεβαίωση για την νομιμότητα και την κανονικότητα των συναλλαγών κιόλας. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούμε πώς, πώς θα γίνει τελικά. Αλλά εάν πάμε προς την ίδια κατεύθυνση νομίζω πως είναι σχεδόν θετική αυτή η τελευταία δήλωση αλλά ας προσπαθήσουμε να μείνουμε έτσι ρεαλιστές και κάπως τεχνοκρατικοί. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό καθόλου. Γιατί είναι καλή η δημοκρατία, αλλά δεν είναι μόνο εκλογές και συζητήσει στην τηλεόραση. Ε, πρέπει να έχει και ουσία και κάποιος πρέπει να διασφαλίσει και αυτή την ουσία. Και αυτό είναι το δικό μας το έργο εδώ πέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ακρόαση αυτή, η οποία πήρε αρκετό χρόνο. Περνάμε στο τελευταίο θέμα. Η ειδική έκθεση 13-2009 για τις εκτελεστικές υπηρεσίες, τις εξωτερικές εκτελεστικές υπηρεσίες, οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου, τον δικαστή Βάρη, να είναι πάρα πολύ σύντομος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Ζητώ συγγνώμη βέβαια για όποιες παραλήψεις ή κενά θα έχει η παρουσίασή μου. και θα σας στείλω φυσικά και την πλήρη έκθεση. Η ειδική έκθεση την οποία λοιπόν έχω την τιμή να σας παρουσιάσω έχει σαν στόχο να εξετάσει αν η εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση ορισμένων προγραμμάτων δαπανών σε σχέση με τις αποκεντρωμένες ή εξωτερικές υπηρεσίες είναι μια ουσιαστική θετική επιλογή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας Κατά τη διάρκεια της μελέτης ανταποκρίνομαι ουσιαστικά ε, σε ένα σαφές αίτημα το οποίο διατύπωσε το Κοινοβούλιο εδώ και λίγο καιρό. Το θέμα είναι να δούμε αν πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τις εξωτερικές υπηρεσίες, οι αποφάσεις αυτές έχουν λάβει υπόψη τους την πραγματική ανάλυση ε, των αναγκών και των ε, πραγματικών ε, ωφελημάτων, αν θα έλεγα, από μια νέα τέτοια λειτουργία. Να δούμε αν μπορούν να οδηγήσουν σε μια εξοικονόμηση δαπανών επίσης και αν μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των εξωτερικών οργάνων. Και ταυτόχρονα αν έχει κατανοήσει σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ρόλο τον ελεγκτικό της λειτουργίας των εξωτερικών υπηρεσιών αυτών μετά από την ακρόαση που είχε, από την ελεγκτική προσπάθεια που είχε γίνει στα πλαίσια των περισσότερων από, αυτών, από αυτές τις εξωτερικές οργανώσεις. Δίδεται η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεντρωθεί στον πυρήνα της λειτουργίας της, το core business, δηλαδή την στρατηγική καταγραφή των αναγκών και την διαμόρφωση των πολιτικών δίνοντάς της την εντύπωση, την δυνατότητα μάλλον να εκχωρεί κάποιες από τις αρμοδιότητες αυτές. Έχει διαπιστώσει λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο ότι αυτές οι εκτελεστικές υπηρεσίες λειτουργήσαν και προσπαθώντας να ικανοποιήσουν σε πρακτικό επίπεδο τις συγκεκριμένες ανάγκες, ιδιαίτερα μετά τη διάλυση των εξωτερικών τεχνικών γραφείων, εκορώντας επίσης και σε εξωτερικές ε, ιδιωτικές υπηρεσίες μερικές φορές τις αρμοδιότητες που είχαν αυτά τα εξωτερικά τεχνικά γραφεία και ταυτόχρονα να προσπαθήσουν να αξιολογήσουν την φύση και τα ειδικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν ε, σε εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων τέτοιου είδους. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα και πιθανώς για την δημιουργία νέων εξωτερικών υπηρεσιών, αξιολογώντας και την καταλληλότητα του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο θα πρέπει να έχουν. Και ξέρετε ότι έχει μεσολαβήσει και ένα screening για τις ανάγκες σε επίπεδο προσωπικού στο τέλος του 2007. Τα θέματα αυτά έχουν συζητηθεί και στη δική σας Επιτροπή σχετικά πρόσφατα και τέθηκε το θέμα ε, ως μη υπάρχουν ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν τίθεται ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αναφέρομαι εδώ στην ανάλυση κόστους και ωφέλους. Ε, των μη οικονομικών παραγόντων όμως. Οι αναλύσεις αυτές περιορίστηκαν στην εξέταση ε, μόνο οικονομικών παραγόντων, παραγόντων κόστους, Και μάλιστα εκεί υπήρχαν και ορισμένα προβλήματα γιατί δεν μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη μας κάποια, κάποια τμήματα του κόστους λειτουργίας και κάποιες μορφές συνεργασίας μεταξύ τους των οργάνων αυτών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα συμπεράσματα λοιπόν είναι ότι η συνεισφορά της ανάλυσης αυτής κόστους-οφέλους για τη δημιουργία των ε, εξωτερικών αυτών γραφείων είναι σχετικά περιορισμένο. Το δεύτερο ερώτημα είναι η οικονομική δικαιούχοι. Η οικονομική δικαιούχοι κατά τη διάρκεια των λειτουργιών αυτών των εξωτερικών εκτελεστικών υπηρεσιών έχουν μεγάλη σημασία. Το 70 περίπου της ε, των εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτές είναι ε, συμβασιούχοι. Αυτό φυσικά είναι μια προφανής εξοικονόμηση χρήματος και το κόστος ε, αμοιβή αυτών των υπαλλήλων είναι το ίμιση του κόστους αμοιβή των μονίμων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με τα ίδια θέματα. Να προσθέσω εδώ ότι από την εξοικονόμηση αυτού του κόστους θα πρέπει να προσθέσουμε βέβαια κάποια επιπλέον κόστη για τη δημιουργία νέων θέσεων λεγόμενων οριζοντίων ε, κάποια κόστη τα οποία θα χαρακτήριζα υποστηρικτικά της λειτουργίας των οργανισμών αυτών. Πράγματι η πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων εξαρτάται και από την ικανότητα του προσωπικού να φέρει πέρα στις συγκεκριμένες αποστολές και από την κατάργηση κάποιων θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων στα πλαίσια της νέας οργάνωσης των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχουμε βέβαια πάρα πολλά στοιχεία σε σχέση με την κατάσταση στο παρελθόν σχετικά με την παραγωγικότητα του προσωπικού. Και δεν έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία για την κατανομή των ρόλων του προσωπικού. Και αυτό δεν έχει επιτρέψει στο ελεγκτικό συνέδριο εξ των να ελέγξει την επαλήθευση των προβλέψεων οι οποίες είχαν γίνει στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει όλα τα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να έχει στη διάθεσή της για το προσωπικό που ασχολείται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στο εσωτερικό της. Σχετικά τώρα με τους λειτουργικούς ή διαχειριστικούς δικαιούχους. Ε, Αυτοί διασφαλίζουν την καλύτερη επίδοση ε, το, στις αυτών των εξωτερικών ε, οργανισμών, εξασφαλίζουν την απλοποίηση των διαδικασιών, εξασφαλίζουν την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και συνεισφέρουν επίσης στην αύξηση της, ε, ε, τη βελτίωση μάλλον της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρωπαϊκό κοινό, στους ευρωπαίους πολίτες. Οι διαδικασίες ε, πρόσληψης υπαλλήλων με ειδικά χαρακτηριστικά απεδείχθη πιο δύσκολη από ό,τι είχε προβλεφθεί και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί επηρέασε αν θέλετε και το χρόνο εκκίνησης λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών. Στα πλαίσια του ελέγχου τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επηρεάζεται αρνητικά από ορισμένου παράγοντες μεταξύ των οποίων το ότι οι αιτήσιες μορφές εργασίας αυτών των εξωτερικών υπηρεσιών λόγω ακριβώς του περίπλοκου χαρακτήρα λειτουργίας τους δεν επιτρέπουν να ελέγξουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει σε σχέση με τα αποτελέσματα. Και καταλήγω στη σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου. Συστήνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τις διαδικασίες εντοπισμού του δυναμικού της εξωτερικοποίησης κάποιων δραστηριοτήτων και τη ζητάμε να λάβει κάποιες νέες αποφάσεις σε σχέση με την διεύρυνση ε, των, του αριθμού των υπηρεσιών αυτών, την αύξηση του αριθμού των υπηρεσιών αυτών. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιώσει και τις διαδικασίες λήψης απόφασης. Θα πρέπει επίσης να δώσει πιο αξιόπιστα στοιχεία σε σχέση με την παραγωγικότητα των εξωτερικών υπηρεσιών αυτών και εκ των υστέρων αλλά και εκ των προτέρων. Θα πρέπει επίσης να εντοπίσουμε και τους παράγοντες επιτυχίας κάποιων τέτοιων εξωτερικών υπηρεσιών και υπάρχουν τέτοιοι, να καταλήξουμε σε πιο αποτελέσματα ικανοποιητικά έτσι ώστε κάποια προγράμματα τα οποία συνεχίζουν να γίνονται αντικείμενο εσωτερικής διαχείρισης να επανεξεταστούν. Θα πρέπει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του ελεγκτικού της ρόλου να θέσει κάποιους νέους στόχους οι οποίοι να έχουν σαν βασικό προσανατολισμό τα αποτελέσματα, την επίτευξη αποτελεσμάτων ίσως να χρησιμοποιήσει για να κρίνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών λιγότερους δείκτες από ό,τι το κάνει τώρα, αλλά δείκτες πιο χαρακτηριστικούς και πιο χρήσιμους. Σας ευχαριστώ για τον σύντομο τρόπο με τον οποίο μας παρουσιάσατε την έκθεσή σας και δίνω το λόγο στην κυρία Χέρτσόγκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πολύ καλή και επίκαιρη ιδέα για την ειδική αυτή έκθεση γιατί όλοι ξέρουμε πως ε, τον να αντικατασταθούν αυτές οι υπηρεσίες από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες ήταν πάρα πολύ σωστό αλλά πρέπει να δούμε και τις εκτελεστικές υπηρεσίες να υπενεμίσω συναδέλφους πως, ε, ε, που πάντα θεωρούν πως έχουν πάρα πολλές υπηρεσίες και απαλλαγές, πως οι εκτελεστικές υπηρεσίες είναι αυτές στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα να εκδώσει απαλλαγή. Οπότε πρέπει να ευχαριστήσουμε εδώ πέρα το ελεγκτικό συνέδριο γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα και για να έχουμε καλύτερο έλεγχο μάλλον θα πρέπει να ζητήσουμε από το Ελληνικό Συνέδριο κάθε 3-5 χρόνια να μας φέρνει εδώ πέρα μια τέτοια ανάλυση για να έχει το Κοινοβούλιο την ευκαιρία να ελέγχει τις εκτελεστικές αυτές υπηρεσίες όχι όπως τις υπόλοιπε, αλλά οπωσδήποτε καλύτερο από τον, δίνει απαλλαγή κομισιών. Επίσης θα ήθελα να πω πως όταν μιλάμε για εκτελεστικές υπηρεσίες μιλάμε για θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εικόνα που δίνουν η μας αφορά όλους μας. Εξάλλου μιλάμε για 32 δισεκατομμύρια που αναλογούν σε αυτές τις υπηρεσίες και για 1.339 υπαλλήλου. Οπότε είναι μεγάλη δουλειά και πρέπει επιγόντω να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες. Κατά τη διάρκεια τη σύνταξη αυτή τη έκθεση ο κύριο Βάρη συνεργάστηκε πάρα πολύ με τον συγητή του Κοινοβουλίου. Συζητήσαμε τα ζητήματα και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ανοιχτή και αποτελεσματική συνεργασία με το Ελληνικό Συνέδριο. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες uh, που αποτέλεσαν αντικείμενο του κυρίου Βάρη. Απλά θα πω κάποια συμπεράσματά μου που μάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, από εμάς έτσι ώστε να ζητήσουμε από την Κομισιόν άλλες απαλλαγές στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα, όπως βλέπουμε από την έκθεση της ε, Κομισιόν, δεν ελέγχονται πλήρως οι δραστηριότητες, γι' αυτό πρέπει να αναπτυχθούν ε, νέοι δείκτες για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα από τις εποπτεύουσες γενικές διευθύνσεις. και βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να αξιολογούμε κυρίως με βάση τις ελλείψεις προσωπικού αλλά τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ άσκησης πολιτικής και εφαρμογής των έργων. Όμως έχουμε την ε, άποψη πως ε, δεν θα πρέπει να συσταθούν νέες υπηρεσίες εκτός εάν προκύψουν νέες αρμοδιότητες κομισιών μέχρι το 2014. Όπως είπε ο κύριος Βάρη, έχουμε εξοικονόμηση κόστους από τη μισθοδοσία, καθώς 75% των υπαλλήλων είναι σύμβασιούχοι και έχουμε εξοικονόμηση κατά 50%, οπότε είναι κάτι το θεσπέσιο αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε πως κάποιες από αυτές δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν να λειτουργούν εγκαίρως, οπότε ποιο το νόημα του να μην μπορεί να ξεκινά γιατί τελικά δεν έχει υπαλλήλους, γιατί δεν μπορούν να τους βρουν και να τους χρηματοδοτήσουν. Άλλες φορές μιλάμε για μήνες, άλλες φορές για χρόνια no at all, uh, like some... και άλλες φορές ε, μιλάμε για το ότι δεν βρίσκουν υπαλλήλους για πολύ καιρό και δεν έχουν ξεκινήσει καν τη λειτουργία τους. Οπωσδήποτε, το βλέπουμε αυτό από τη Σκοπιά, της ε, Γενικής ε, Διεύθυνσης Προσωπικού και βέβαια πρέπει να ξεχνάμε πως αν ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να πάει ε, σε θέση με 50% καλύτερο μισθό δεν θα πάει στις εκτελεστικές υπηρεσίες οπότε δεν ξέρω πρέπει να το δούμε πως απλά χάνουμε χρόνο, χρήμα και την καλή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν λειτουργούν σωστά αυτές οι υπηρεσίες πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται ειδικά καθώς χρειαζόμαστε εξειδικευμένη γνώση και προσωπικό. Νομίζω λοιπόν κύριε Πρόεδρε πως θα τελειώσω εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία με το Ελληνικό Συνέδριο και τους Κιώδης και η Επιτροπή μας παρά το ότι δεν μπορεί να δώσει απαλλαγή πρέπει να βλέπουμε που και που αυτά τα ζητήματα. Οπότε πρέπει να μας ε, δίνει αναφορά το ελεγκτικό συνέδριο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Ο μιλό εκπρόσωπο τη κυρία Συγγήτρια κυρία Ρόλμανερ και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και την κυρία Χέρτσοκ επίση, η οποία πράγματι έχει δείξει πολύ μεγάλη ικανότητα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα των ε, υπηρεσιών. Φυσικά έχουμε πολύ σημαντικούς, ε, σημαντικές επιπτώσεις από την τήρηση των κανόνων, έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες και έχουμε ε, μεγάλη επιβάλληση μισθολογική βεβαίως το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό αλλά έχουμε εντωμεταξύ 40% συμβασιούχους πράγμα το οποίο δημιουργεί σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις ε, και την υποχρέωση να πληρώνουμε με ισότιμο μισθό την ίση εργασία. Άρα θα έλεγα ότι η μορφή, η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί δεν είναι δίκαιη γιατί δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτό το οποίο οφείλουμε να προσφέρουμε. Και αυτό θα ήθελα να γίνουν κάποιες ορθώσει. Ευχαριστώ πολύ, Αγιάλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, οφείλω να ευχαριστώ την κυρία Χέρτσοκ για το σχέδιο έκθεσης οι οργανισμοί που εγώ έχω υπόψη μου, εκτελεστική, κανονιστική, μια εκτελεστική που ασχολείται με τις μεταφορές ιδιαίτερα. Ε, τους γνωρίζω λοιπόν αρκετά καλά. Οφείλω να πω όμως ότι με καταπλήσει η δήλωση ότι αυτοί οι εκτελεστικοί οργανισμοί δεν είναι τίποτε άλλο από ανα, ε, ε, νέο όνομα, εν πάση περιπτώσει, για τις παλιές υπηρεσίες που δεν θα θέλαμε να επανέλθουν με αυτή τη μορφή. Γι' αυτό λοιπόν διαρωτώ με εάν μπορούμε να καταλήξουμε στα αποτελέσματα, στα συμπεράσματα στα οποία ε, μας καθοδηγείτε εσείς. Το θέμα δεν είναι αν θα έχουμε πιο φθηνό προσωπικό ή όχι, αλλά αν θα έχουμε επαρκή ευελιξία στο προσωπικό μας, ώστε ή μάλλον στις ε, συνθήκες που προσφέρουμε ώστε να εξασφαλίσουμε και το καλύτερο δυνατό προσωπικό. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι ικανότατοι αλλά δεν έρχονται σε εμά διότι δεν τους προσφέρουμε αρκετά, καλά, ε, αρκετά καλές προοπτικές ε, οι συνθήκες. Και εδώ έχουμε να κάνουμε συμβάσεις που είναι μερικές φορές επτά είναι ε, παράταση. Ερωτώ λοιπόν και για τον κύριο Ευάρη αν αυτό ισχύει για όλους τους οργανισμούς αφενός, αφετέρου δε, εάν η κατάσταση είναι ομοιόμορφη ε, παντού, διότι η εκτελεστική, ο εκτελεστικός οργανισμός για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, παραδείγματι, δεν έχει τέτοιες συνθήκες και αυτό ισχύει. Γενικά τα προβλήματα που έχουν οι συμβασιούχοι είναι κοινά και εδώ στο Κοινοβούλιο και στις Επιτροπές Συμβασιούχοι και γενικά όπου υπάρχουν συμβάσεις και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή μαζί με την κυρία Κρέσλη, θα συμφωνήσω και εγώ ότι χρειάζεται δηλαδή να δούμε αυτά τα ζητήματα της αντίστοιχης αμοιβή. Ε, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίω ότι θα πρέπει ο στόχος τελικά να είναι ένα χαμηλότερη αμοιβή που δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο κύριος Βάρη για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Χέρτσογκ όπως επίσης και τις ε, δύο άλλες συναδέλφους της για τα καλά της λόγια, την κυρία Γκρέσλα και την κυρία Γιάλα. Σχετικά με τα θέματα προσωπικού. Νομίζω ότι τα θέματα αυτά τίθενται με τον ίδιο τρόπο για όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες. Τα κριτήρια πρόσληψης είναι τα ίδια για όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες. Και αν μου επιτρέπει ο Πρόεδρος, μιας και εξετίμησε την συντομία με την οποία, με την οποία παρουσίασα, θα ήθελα πέντε λεπτά να μου δώσει για να επιστήσω την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παράγραφο 50 γιατί επαναλαμβάνω ότι το θέμα του προσωπικού είναι ένα από τα κεντρικά θέματα της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Σας διαβάζω την παράγραφο αυτή. Λέγεται ότι η πρόσληψη του προσωπικού οι ειδικέ ικανότητες είναι μια διαδικασία η οποία πήρε πολύ περισσότερο χρόνο από όσοι υπολογίζαμε, από όσον υπολογίζαμε. Και η κάλυψη των κενών του οργανογράμματος ακολουθεί τους κανονικούς κανόνες πρόσληψης που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της συγκεκριμένη Γενικής Διεύθυνσης. Οι προσλήψεις στις εξωτερικές υπηρεσίες ε, γίνονται κυρίως ή μάλλον στις μόνιμες υπηρεσίες γίνονται σε χαμηλού βαθμού υπαλλήλου, ενώ ε, στις εξωτερικές υπηρεσίες επιζητείται για τους συμβασιούχους μια μεγάλη επαγγελματική πείρα παρότι προτείνονται επαναλαμβανόμενες συμβάσεις αντίθετα με τις τριετή συμβάσεις οι οποίες συνήθως χορηγούνται σε ε, συμβασιούχους οι οποίοι προσλαμβάνονται από τις κεντρικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν θέλετε να προετοιμάσω περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με όλα αυτά. Είμαι στην ε, διάθεσή σας, θα βρείτε κάποια από αυτά που ζητάτε στο γραπτό κείμενο. Καλώς, τελειώσαμε. Υπάρχουν κάποια πρακτικά θέματα στα διάφορα. Α, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει κάτι να προσθέσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια μάλλον για την έκθεση αυτή, την οποία έχουμε μελετήσει πολύ προσεκτικά, την γνωρίζουμε καλά και κυρίω για τι πτυχέ τη απαλλαγή. Δεν θέλω να υπενθυμίσω στου εκτελεστικού οργανισμού. Υπάρχει πολύ μικρό λειτουργικό προπολογισμό επιδοτήσει, για τον οποίο δίνει χωριστή απαλλαγή το Κοινοβούλιο είναι ένας τεράστιος λειτουργικός προϋπολογισμός για τον οποίο είναι ε, εντολοδόχος της Επιτροπής ε, ο εκτελεστικό οργανισμός. Και τα πάντα υπάγονται στην απαλλαγή πάλι του Κοινοβουλίου μέσω της απαλλαγής στην Επιτροπή. Ε, για το προσωπικό. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε το αντικείμενο της συζήτηση. Δεν μπορείτε αυτή μια να μας λέτε ότι πρέπει να κάνουμε οικονομίες και από την άλλη να πρέπει να πληρώνουμε τα ίδια. Είναι ζήτημα οικονομικών επιλογών, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, πολιτικά ευαίσθητο, είναι εγγεγραμμένο στη συνθήκη, στο κανο... καταστατικό των υπαλλήλων, στον κανονισμό των υπαλλήλων και έχουμε αυτή τη στιγμή υπαλλήλου που δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι σε ορισμένε περιπτώσει. Συμβασιούχοι στου εκτελεστικού οργανισμού κοστίζουν λιγότερο. Αυτό είναι πολιτική βούληση που οδήγησε στη μεταρρύθμιση, που είναι μέσα στο κανονισμό υπαλληλική κατάσταση, που έχει να κάνει με τη διαχείριση των ανθρωπινών πόρων στην Επιτροπή και δεν είναι ένα μεμονωμένο ζήτημα που σχετίζεται με του εκτελεστικού οργανισμού. 5.000 είναι συμβασιούχοι στι υπηρεσίε Επιτροπή και 1.000 εξ αυτών ε, ανήκουν στου εκτελεστικού οργανισμού. μην μπερδεύουμε λοιπόν, μην συγχαίουμε το αντικείμενο της συζήτηση. Εδώ βρισκόμαστε στην, ε, στον πυρήνα τον ίδιο της, επιτροπής, της πολιτικής επιλογής ως προς τη δημοσιοϊπαλληλική κατάσταση. Είναι τεράστιο το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει αν αλλάξουν κάποια από τα ζητήματα, οικονομικό πρόβλημα. Γιατί άκουσα με προσοχή τα όσα υπόθηκαν. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στα διάφορα λοιπόν υπάρχουν τρία θέματα. Το πρώτο σας το είχα υποβάλει, το είχαμε συζητήσει με τη γραμματεία, για να χρησιμοποιήσουμε τις δύο ημερομηνίες, 22 και 23 Φεβρουαρίου, για να συναντηθούμε με τον Σεμέτα. Θα έχει επιβεβαιωθεί ο Σεμέτα τότε και θα ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τα θέματα τα οποία συζητήσαμε σήμερα, εφόσον συμφωνείτε. Ο κύριος Σεμέτα είπε ότι και ο Μπράουν θα είναι διαθέσιμος. Ένα άλλο θέμα, εφόσον συμφωνείτε, θα πρέπει να προβλέψουμε μία συνάντηση των συντονιστών μετά από την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Μία πάρα πολύ σημαντική γνωμοδότηση η οποία δημιουργεί θα έλεγα ένα θέμα στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα. Ένα τρίτο κατεπήγον θα πρέπει να αποφασίσουμε αν το Κοινοβούλιο θα πρέπει, σε σχέση με, θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με την προσφυγή επί παραβάση εις βάρος της Γερμανίας σε σχέση με το ΦΠΑ. Κύριε Ανδρέας, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στα πρακτικά της, ε, του Δεκεμβρίου, 2 και 3 Δεκεμβρίου, χωρίς να θέλω να προτείνω τροποποίηση. Θα ήθελα να επισημάνω το σημείο 8 8Γ επανέρχεται προς συζήτηση, αφορά την ε, διοικηστική μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε όσους ε, καταγγέλουν παρατυπίες ή διαφθορά. Και θα ήθελα επίσης να ζητήσω μια καλύτερη διαχείριση του χρόνου για τους ομιλητές, Πρόεδρε, διότι δεν νομίζω ότι είναι πολύ ισορροπημένη η κατανομή του χρόνου και θα έπρεπε από την αρχή να έχετε περισσότερη, να έχετε προσέξει περισσότερο. Κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε περαιτέρω προσφυγές και να λάβω και εγώ το λόγο. Η επόμενη συνάντηση είναι στις 22 Φεβρουαρίου στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας.